συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη του στόχου τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Άστον. Ευχαριστούμε κύριε Άστον. Έχουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν για την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης από την Ευρώπη των Δημοκρατιών και των Ελευθεριών, από τους Πράσινους στην Ενωτική Αριστερά, άλλοι από τους Φιλελεύθερους, από το ΕΛΚ επιπλέον και κλείνει η συζήτηση με αυτή την ανακοίνωση. Η ψήφιση θα διαξαχθεί αύριο το μεσημέρι, 12.00. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση των συναδέλφων κυρίων Μπροκ και Γκουαλτιέρη για την ε, <clears throat> μεταρρύθμιση και λειτουργία της, ε, Επιτροπής, ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα λάβει τον λόγο πρώτος ο κύριος Μπρόκος, εισηγητής επ' αυτού θα παρέμβει ε, για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ κύριε Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωποι, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι, στη Μαδρίτη τότε καταλήξαμε στο παρελθόν σε μια συμφωνία όπου το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και είπατε εκπρόσωπο ε, συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, ε, Δράσης που ακριβώς θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Θα πρέπει οι ικανότητες και το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ικανότητες και το δυναμικό του Συμβουλίου, χωρίς την αλλαγή αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, να συγκλίνουν σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στα εξωτερικά θέματα. Και οι αναγκαίες συνέργειες πρέπει να επιτευχθούν, ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε όπως δεν μπορούσαμε στο παρελθόν και θα πρέπει να πούμε μπορεί το ποτήρι να είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο όμως είναι μισογεμάτο περισσότερο. Κατά τη διάρκεια αυτού, του χρονικού διαστήματος πετύχαμε πάρα πολλά και βαρώνει άστον σε μια ολόκληρη σειρά τομέων, ένα παράδειγμα είναι η Σερβία και το Κωσυφοπέδιο. καταφέραμε πολλά σημαντικά πράγματα. Βλέπω όμως ότι ο κινητήρας δεν λειτουργεί χωρίς προβλήματα πολλές φορές και ίσως επειδή ο ρόλος της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι εκείνος ο οποίος ε, εκφράζει αυτή την, αυτό τον κινητήρα. Πρέπει να είναι σαφές ότι η πολιτική γειτονία είναι μια πολιτική που μπορεί να δράσει μέσα στο πλαίσιο των μέσων και πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι στον τομέα όμως και του Συμβουλίου τα πράγματα δεν προχωρούν όπως θα έπρεπε. Στο Μάλι αποφασίστηκε τον Οκτώβριο να αποστείλουμε μια αποστολή κατάρτισης προς τους ε, ε, στρατιωτικούς του Μάλι και μέχρι ε, μερικούς μήνες πριν δεν είχε γίνει τίποτα μέχρι τον Ιανουάριο. Η διαθροτική συνεργασία δεν προήχθη και σε σχέση με την προαγωγή των battle groups, ε, των ομάδων μάχης. Πρέπει να προβληματιστούμε πώς μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις και να υπάρξουν κίνητρα ώστε η ύπατος ε, εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μπορεί να οδηγήσει στην λήψη σωστών πρωτοβουλειών που θα συνοδεύονται και από τι αναγκαίε πρωτοβουλίες του Συμβουλίου. Εσωτερικός μηχανισμός δηλαδή να ενισχυθεί σε σχέση με το δυναμικό που έχουμε να παρεμβαίνουμε και να δρούμε. Αυτό πρέπει να γίνει λοιπόν και να διασφαλιστεί με το ότι θα αποσαφηνίσουμε με σαφήνεια ότι αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να είναι υπόθεση κρατών μελών. Και αν δούμε την χώρα την οποία γνωρίζω καλύτερα, που πολλές φορές θέλουν μέσω οι εκπρόσωποι αυτής της χώρας να δούμε μέσω των πρέσβεων τον Ιούνιο του 2013 θα μπορούν μέσω των κανονικών διαδικασιών να ε, λειτουργούμε και να δρούμε. Δεν είναι δυνατόν 30% ε, να ε, προσλαμβάνονται και να δρούμε μόνο από πλευρά των κρατών μελών. Πρέπει όλα να γίνονται με τον ίδιο τρόπο και ταυτόχρονα και να υπάρχει και έλεγχος, να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε γέφυρες και να είμαστε αποτελεσματικοί και όσον αφορά τις πρεσβείες μας. Και το θέμα του ελέγχου επίσης σημαντικό. Η δραστηριότητά μας πρέπει να διασφαλιστεί και η αποτελεσματικότητά μας όμως. Και εξακολουθούμε να έχουμε δυσκολίες όσον αφορά το reporting, τις αναφορές προς λογοδότηση και αξιολόγηση και την διαβίβαση συστάσεων και κατευθύνσεων. Πρέπει να είναι σαφές, άσχετα αν είναι το διακυβερνητικό τμήμα συνεργασίας ή το κοινωνικό τμήμα, ότι μόνο μέσω αυτών των πρεσβειών θα μπορούμε να δρούμε ώστε να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν και επινοήθηκαν ώστε να μπορούμε από κοινού κοινοτικά να δρούμε, συνεκτικά και όχι εμβαλωματικά. Να μπορούμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό η εξωτερική υπηρεσία Βαρώνη Άστον πρέπει να μπορεί να δίνει βοήθεια και να υπάρχει αυτή η συνεργασία και αυτή η συνέργεια. Θέλουμε ε, σε τακτά διαστήματα να μπορεί να υπάρχει μια αξιολόγηση. Ε, αποκινούμε τον κύριο Γουαλτιέρη, δίνουμε προτάσεις και κίνητρα για αυτή την, προς αυτή την κατεύθυνση, για αυτή τη δράση και ελπίζουμε ότι θα ξανασυναντηθούμε το φθινόπωρο και θα μας πείτε ποια συμπεράσματα έχετε συναγάγει και ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις ώστε στη συνέχεια να έχουμε μια σημαντική αποτελεσματική εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπροκ. Κύριε Μπροκ, προσέξτε, με ακούτε. Γνωρίζετε ότι Είσαστε παλαιός κοινοβουλευτικός, έχετε έξι λεπτά για να παρέμβετε κανονικά. τέσσερα και δύο για να ολοκληρώσετε. Αλλά όταν έχετε χρησιμοποιήσει πέντε στην κύρια παρέμβασή σας, απομένει ένα λεπτό μετά για να ολοκληρώσετε. Θα έχετε ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Και τώρα θα έχει τον λόγο ο κύριος Γκουαλτιέρη με την ίδια επισήμανση προς εκείνον προτού ξεκινήσει για να γνωρίζει πώς θα κατανείμει το χρόνο του όπως θεωρεί πιο σκόπιμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε το ψήφισμα, η έκθεση μάλι που θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο θέλει να συνδράμει με επικοδομητικό τρόπο στην όλη θεώρηση. Ε, και αυτό βάρει μιας ε, αποτίμηση των πρώτων ετών δραστηριοτήτων που εντόμισε προβλήματα και όρια και ταυτόχρονα αναγνωρίζει και αξιοσημείωτες πρόοδους ε, που σημειώθηκαν σε λίγα χρόνια. Όταν θέλαμε να επικυρώσουμε τις υπηρεσίες του 2010 ξέραμε ότι θα έπρεπε να ενταχθεί στη δομή να ενταχθούν στη δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου υπάλληλοι των κρατών μελών και αυτό ήταν κάτι φιλόδοξο. Το Κοινοβούλιο παρετείται το αίτημά του να μπει η υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει μια ευρύτερη υπηρεσία που να μπορεί να πηγαίνει την πολιτική ασφάλεια και κοινή άμυνα προ την πολιτική την αναπτυξιακή και ταυτόχρονα να είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπόκειται σε έναν επαρκή έλεγχο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ο στόχο επετεύχθη τότε και πραγματοποίησαμε, υλοποίησαμε μια υπηρεσία που πιστεύω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό, που έχει ευρύτερε αρμοδιότητε από αυτέ που ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι θα ήθελε το Συμβούλιο και θα υπόκειται σε έναν έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγαλύτερο από αυτό που ήθελαν και οι δύο, τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Αυτό προσφέρει στην Ένωση ένα εξαιρετικό εργαλείο για να πραγματοποιήσει μια σφαιρική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική. Να ευνοήσει μια σύμπραξη μεταξύ των διαφόρων εργαλείων που διαθέτει η Ευρώπη στην εξωτερική τη δράση και που συνάδουν με μια φιλοσοφία για την εξωτερική πολιτική που παίζει κυρίαρχο ρόλο όσον αφορά τη χρήση τη ήπια δύναμη, soft power, δηλαδή συνένεση, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη των λαών, χωρί ταυτόχρονα να παρετούμεθα από τα στατιωτικά μέσα για τη διαχείριση των κρίσεων και το στόχο να οικοδομήσουμε μια κοινή άμυνα. Οι προτάσει που παρουσιάζουμε σήμερα δεν θέλουν να αλλάξουν τη βάση που καθορίστηκε το 2010 και αντίθετα παγιώνουν ε, τη σωστή αυτή βάση. Η δική μα έκθεση προτείνει όμω να εντοπιστούν τα προβλήματα που δεν επιτρέπουν στην υπηρεσία αυτή να εκφραστεί όπως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δυναμικό της. Εντοπίζει κάποιες ενδεχόμενες λύσεις που θεωρούμε ότι είναι συνεκτικές και ταιριάζουν με τη βασική κατεύθυνση που επελέγει το 2010 και επιδιώχτηκε αυτά τα χρόνια. Δεν επαναλαμβάνω τις προτάσεις που ήδη ανέφερε ο συνάδελφος Μπρόκ. Ε, λοιπόν, ε, το, ε, λοιπόν, δεν νομίζω υπάρχουν αμφιβολίες για τους στόχους. Εξορθολογισμός της δομής. Θέλουμε την ενίσχυση του ρόλου της αντιπροέδρου, του αντιπροέδρου ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη ΣΥΠΑ τη εκπροσώπου, ποιε είναι οι δομέ για τη χείριση των κρίσεων, θέλουμε ενίσχυση του ρόλου των επικεφαλή των αντιπροσωπιών, θέλουμε πλήρη πολιτικό έλεγχο από πλευρά του Κοινοβουλίου, θέλουμε αυτονομία των διαδικασιών τη προσλήψεω ε, όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Είναι λογικέ προτάσει πιστεύουμε, κάποιε θα μπορούσαν να υλοποιηθούν επί τη βάση τη αποφάσεω που ήδη ισχύει, ενώ άλλε αλλαγέ θα πετέσουν μια τέτοια τροποποίηση, αναθεώρηση τη απόφαση και γι' αυτό ζητούμε να να συμμετάσχει πλήρω στο Κοινοβούλιο παρόμοια όπως ε, παρενέβη και το 2010 για να αλλάξουν αυτά. Λοιπόν, μέσω του διαλόγου ε, έχω την πεποίθηση ότι μαζί σας κυρία Πατιακπρόσωπος θα έχουμε καρποφόρο διάλογο και ότι ε, η εξωτερική αυτή υπηρεσία εξωτερική δράση θα δώσει ένα καλύτερο εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει μια πολιτική εξωτερική που θα ανταποκρίνεται και στι ευθύνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στι φιλοδοξίε τη. Σα ευχαριστούμε κύριε Γκουατιέρη. Θα λάβει τον λόγο η κυρία Άστον για να απαντήσει στους δύο εισηγητές αυτής της τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι μια ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς τον κύριο Μπροκ ε, και τον κύριο Γκουαλτιέρη για την εξισορροπημένη έκθεσή τους. Μαζί με τον Φερ Χωστάτη είσαστε οι ιδρυτές, υποστηρικτές της Συμφωνίας της Μαδρίτης που ε, που υπήρξε σημαντική για τη δημιουργία της υπηρεσίας και σας ευχαριστώ για αυτά που αναφέρετε στην έκθεση. Η ιδέα μας ήταν να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία ευρωπαϊκή του 21ου αιώνα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και να κάνουμε κάτι παραπάνω από τα Υπουργεία Εξωτερικών, διότι έχουμε και στοιχεία ανάπτυξης και άμυνας. Η ισχύ μας στηρίζεται στην ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις κρίσεις με πολύ ευρύτερο τρόπο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο για την ε, ε, ανάπτυξη, για την, ε, ανάπτυξη την ασφάλεια, την προστασία των ανθρώπων κλπ. Δυόμιση χρόνια μετά τη διίδρυση της υπηρεσίας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική υπηρεσία η οποία προσελκύει τους καλύτερους υπαλλήλους και διπλωμάτες από όλη την Ευρώπη. Ρόλος της είναι να προσφέρει, να προσφέρει, παρέχει ε, νοσιακές πολιτικές. Τώρα που βλέπουμε τις αλλαγές τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε. Για μένα τρία είναι τα σημαντικά στοιχεία στα οποία θέλω να εστιαστώ. Πρώτον, η γειτονιά μας, η γειτονία μας. Όταν μου ζήτησαν να αναλάβω αυτά τα καθήκοντα, είπα ότι πρέπει να, να ορίσω, πρέπει να ορίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που μπορούμε να κάνουμε στη δική μας γειτονιά. Ε, μπορούμε να ασκήσουμε τεράστια επιρροή για να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τις μεταβολές στη γειτονιά μας που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Δεύτερον, η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η συγχώνευση τριών ιδιωτήτων ε, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τα διάφορα μέσα που διαθέτουμε, να υποστηρίξουμε το κράτος δικαίου, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την αναπτυξιακή μας βοήθεια, την διπλωματία μας ε, δράσεις που αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα αλλά και τους, ε, τα αίτια που οδηγούν σε αυτά τα συμπτώματα και έχουμε μια κρίσιμη μάζα, τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διεθνώς. Συλλογικά μπορούμε να, πετύχουμε, να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα που μονομένα τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να κάνουν. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, υποστηρίξει τις προσπάθειές μας στο Ιράν, στην Σομαλία, στο Κόσοβο πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την ικανότητά μας, ε, να ε, ε, παρεμβαίνουμε και να έχουμε δράση σε όλους αυτούς τους τομείς. Οι φιλοδοξίες μας είναι μεγάλες και σας ευχαριστώ για την έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Να γίνουμε καλύτεροι, να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι στην εφαρμογή των διαφόρων διαδικασιών και για τον ρόλο του Αντιπροέδρου της Επιτροπής που θα εξασφαλίσει όλες τις εκτερικές σχέσεις πολιτικής μας μας. Με ενθαρρύνουν οι, αντιδράσεις των, θετικές αντιδράσεις των κρατών μελών που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Η επιτυχία της υπηρεσίας μας στηρίζεται στη δυνατότητα να φέρνουμε κοντά τις διάφορες, ε, τα διάφορα όργανα ενώ θα περιορίζουμε ταυτόχρονα για, αποτελεσματικά ε, να πετυχαίνουμε καλά αποτελέσματα περιορίζοντας ταυτόχρονα το κόστος. Θέλω να υπογραμμίσω τι ε, ε, ε, ενεργεί ε, σωστά, τι εφαρμόζεται σωστά, αλλά τι άλλο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Θα υπάρξουν αλλαγές και κάποιες προσαρμογές που θα απαιτηθούν μετά τη λήξη της θητείας. Αυτές οι συστάσεις θα έχουν σκοπό να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μας. Δεν πρέπει ωστόσο να έχουμε αυταπάτη. Πρέπει να θεωρήσουμε να θεωρήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις με βάση την πολιτική βούληση και τη συμφωνία όλων των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε όμως τη σύριξη των κρατών μελών για να ε, προσφέρει η υπηρεσία μας ό,τι το καλύτερο μπορεί. Πρέπει να ε, πρέπει να προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε τη συνένεση ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη, συνεργαζόμενοι πιο στενά με και με την Επιτροπή η υπηρεσία με υποστηρίζει στη θέση του ΥΠΑ του εκπροσώπου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής και, με τον, για αυτό τον και, σαν αποτέλεσμα θα μπορέσουμε να κάνουμε τον συντονισμό το που ζητάει η έκθεση. Η συμφωνία που έχουμε για την πολιτική λογοδοσία έχει, έχει προσφέρει μεγάλες... Ε, μεγάλη σημαντική εξέλιξη. Ε, έχουν γίνει αλλαγές στον τρόπο που γίνεται ο διορισμός των επικεφαλής των αντιπροσωπιών, στο, κάτι στο οποίο αποδίδουμε όλοι μεγάλη σημασία. Εξαιρετική συνεργασία σε ό,τι αφορά τις αποστολές ε, εποπτείας, επιτήρησης των εκλογών. Εντατικότερος διάλογος σε όλα τα επίπεδα ε, ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές που απαιτούν την, ε, την ανακοίνωση ευαίσθητων πληροφοριών, την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, το 2012 είχαμε πάνω από 200 εκδηλώσεις και συγχαίρω τους αρχηγούς των αντιπροσωπιών που, έχουν, που βοηθάνε τόσο πολύ στην οργάνωση των επισκέψεων υψηλών αξιωματούχων. Στην ίδια την έκθεση θέλω να αναφερθώ σε τρεις συγκεκριμένους τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η συνεργασία με την Επιτροπή. Τους, επίσης, πολλά ερωτήματα έχουν τεθεί για τη συνεργασία μεταξύ υπηρεσίας και Επιτροπής και αναφέρθηκαν στις αρχικές δηλώσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι κάποιες φορές υποτιμάμε, υποτιμούμε την πρόοδο που έχει επιτευθεί προτείνοντας λύσεις στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ανατρέχοντας πίσω δεν ξέρω αν είχαμε υποτιμήσει το εύρος αυτής της εργασίας αλλά σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο εξακολουθούμε να συζητούμε με την Επιτροπή συμπεριλαμβανομένου και του θέματος να χρησιμοποιούμε περισσότερο την ομάδα της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι γίνεται ήδη πολύ εντατική δουλειά με τους Επιτρόπους για τη Γεωργία, τον Επίτροπο Γεωργίας ο οποίος θα παίξει ζωτικό, ζωτικό ρόλο τον Νοέμβριο, Σίλια Μάντσρομ, Νέλα Κρούς, για τα θέματα της προστασίας του κυβερνοχώρου. Ο Επίτροπος που φροντίζει, που φροντίζει για το, το, το, το τομέα των επιχειρήσεων, ο Μισελ Μπαρνιέ και εγώ, ε, συμμετέχουμε στις συζητήσεις για το, την αμυντική βιομηχανία. Επίσης, η επιτροπή ε, αυτά όλα, αυτά που, την υποστήριξη που είχαμε από τους επιτρόπους για το θέμα της Συρίας. Αλλά βεβαίως είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που υπογραμμίζεται τη σημασία της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην, στους διάφορους στόχους της πολιτικής. Για το δεύτερο θέμα συμφωνώ με την ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια για το θέμα της ανάθεσης, ανάθεσης αρμοδιοτήτων Σύμφωνα με την έκθεσή σας πιστεύω ότι πρέπει με πιο διαρθρωμένο τρόπο να αναθέτουμε στους επιτρόπους ορισμένες δραστηριότητες και να προχωρήσουμε πιο πέρα από ό,τι έχουμε ήδη φτάσει εντέλλοντας συγκεκριμένες αποστολές σε υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών ώστε να δώσουμε μια μεγαλύτερη όθηση ε, και μεγαλύτερη αναγνώριση στην θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομάδες ε, υπουργών των διαφόρων κρατών μελών θα είναι πολύ σημαντικό να κάνουν επισκέψεις σε διάφορες χώρες. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Χαιρετίζω την έμφαση που δίνεται στις ε, πολιτικές και τις στρατιωτικές μας αποστολές. Ε, στην Πριστίνα, στο Μογκαντίσου, στην Καμπούλ, στην Βαγδάτη και αλλού. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις σας για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα της λήψης αποφάσεων και την ενσωμάτωση των αρμοδίων υπηρεσιών στις υπάρχουσες δομές. Θέλουμε να απλουστεύσουν τις διαδικασίες σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτό θα είναι κάτι το πολύ σημαντικό καθώς προετοιμαζόμαστε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης πρέπει να προσδιορίσουμε καλύτερα τις εσωτερικές δομές δεδομένης της οικονομικής κατάστασης. Για τον προπολογισμό του 2014 θα ζητήσω να μειωθούν οι ανώτατες θέσεις και πιστεύω ότι θα υπάρχει δυνατότητα να, γίνει, να περιοριστούν ακόμα περισσότερα περισσότερες θέσεις. Βεβαίως στην Ευρω... υπολογίζω, υπολογίζω στην συμβολή των κρατών μελών. Πραγματικά, πραγματικά είμαι ιδιαίτερα τυχερή για τους συνεργάτες ε, που με πλαισιώνουν και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για όλη τη σκληρή δουλειά που προσέφεραν τα τρία τελευταία χρόνια. Η ετήσια έκθεση που θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο θα δείξει ότι έχουμε σημειώσει σημαντικούς, σημαντικές πρόοδους σε σχέση με όλα τα κράτη-μέλη και σε ό,τι αφορά την θέση των γυναικών μέσα στις αντιπροσωπείες. 18% ε, του προσωπικού ε, είναι οι γυναίκες που πλησιάζει πάρα πολύ στο 20% που είχαμε ορίσει. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν επίσης την παρουσία ε, ε, αξιωματούχων που έχουν μεταφερθεί σε άλλες χώρες από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Το θέμα της ισότητας ε, μεταξύ των δύο φύλων είναι αποτελεί προτεραιότητα. Σήμερα έχουμε 24 γυναίκες, μια αύξηση πάνω του 100% και έχουν ήδη διοριστεί το 2013 τέσσερις γυναίκες αντιπροσωπείε. Ο Σμιτ ο πολιτικός διευθυντής μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει την ένταξη περισσότερων γυναικών στην υπηρεσία μας. Επίση, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο στόχο του ενό τρίτου για τι προσλήψει των διπλωματών και των μονίμων υπαλλήλων. Βεβαίω χρειάζομαστε μια πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που να προσελκύει ε, τους πολλούς ενδιαφερόμενους συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εργάζονται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Θα αρχίσουν να θα δημοσιευθούν οι κενές θέσεις απασχόλησης στο Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα σήμερα με την απόφαση που έχει ληφθεί και σε ό,τι αφορά επίσης και τους διπλωμάτες από την Κροατία. Βεβαίως θα θέλαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα αλλά μας περιορίζουν ε, οι οικονομικές μας δυνατότητα. Ορισμένοι πόροι κληρονομήθηκαν από το Συμβούλιο και την Επιτροπή και στηριζόμαστε στην Επιτροπή για υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό. Αποφεύγουμε τις επικαλύψεις, προσπαθούμε να οργανώσουμε καλύτερα τα πράγματα στις Βρυξέλλες και θέλουμε να παραμείνουμε, να, παραμείνουμε, να παραμείνει, να συνεχιστεί η παρουσία μας σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Αντιπροσωπείες, αναφέρουμε σε αντιπροσωπείες της Λιβύης και του Μιανμάρ. 30 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την Καβούλ, τη Λιβύα και άλλε χώρε υψηλού κινδύνου. Είμαι πεπισμένο ότι πρέπει να μετατρέψουμε του όρου του προπολογισμού των κρατών μελών για να δούμε ποιε είναι οι δυνατότητε για ε, οικονομίες ε, καθώς θα συνεχίζεται η πρόοδος μας με διάφορες ρυθμίσεις θα συνεργαζόμαστε πιο στενά Η πόροι είναι το στοιχείο κλειδί για την ε, αναδιοργάνωση οποιασδήποτε δραστηριότητες. Υπάρχουν τομείς στους οποίους ακόμα δεν έχουμε αποκτήσει αρκετή εμπειρία. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να περάσει χρόνος. Δεν μπορεί να γίνει μία, εν μία νυχτή. Όπως σας είπα, περάσαμε από το να μην έχουμε καθόλου υπηρεσία σε μία αποτελεσματική, εξαιρετική υπηρεσία. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να ανταποκριθούμε στους συλλογικούς, ε, στις συλλογικές προκλήσεις και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Άστον. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Νεϊνσκι εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών της Ευρωβουλής. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Μπρόκ, αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Τα τελευταία δύο χρόνια ασχοληθήκαμε με τη δομή, τη διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τώρα είναι η χρονική στιγμή να εξετάσουμε την μελλοντική ανάπτυξη και μετεξέλιξη αυτής της υπηρεσίας ως τμήματος της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι η κατανομή και η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών πρέπει να εξαρτάται από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης. Μόνο με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας στην εξωτερική πολιτική της ε, εξωτερικής δράσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο το δυναμικό μας και τα κονδύλια. Δεδομένων των περικοπών και της εξοικονόμησης που είναι αναγκαία στοιχεία, πιστεύω ότι η εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα υπουργεία Υπουργεία Εξωτερικών των κρατών μελών και όσον αφορά και την ανταλλαγή δυνατοτήτων και πειρασμών. Έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ενιαία θα δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι ευρωπαϊκέ προτεραιότητε θα εφαρμόζονται και θα υλοποιούνται. Στο τέλο τέλο, ζητώ από την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να διασφαλίσει την γεωγραφική ισορροπία ώστε να ε, χρησιμοποιούνται περισσότεροι υπάλληλοι και στελέχοι από τα κεντροανατολικά κράτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Άστον για τις προσπάθειες υπέρ της εκπροσώπησης των γυναικών στην υπηρεσία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ε, ρητορική άσκηση θεσμικού χαρακτήρα αυτή η συζήτηση. Είναι ο προβληματισμός μας για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Νέσκι. Δεν βλέπω στο έδρανό του τον κύριο Κάλφιν που έπρεπε τώρα να παρέμβει εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ελπίζουμε ότι θα προσέλθει κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Περνάμε στους αγορητές τώρα, που θα παρέμβουν εξ ονόματος των κοινοβουλευτικών τους ομάδων. Πρώτα απ' όλα για δύο λεπτά θα παρέμβει ο κύριος Άλαφράνκα, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αυτή η σύσταση και δράτω με τις ευκαιρίες για να συγχαρώ τους εισηγητές, τον συνάδελφο κύριο Μπρόκ και τον συνάδελφο Γκουαλτιέρη, βρίσκεται, εντάσσεται στο στόχο και την εξυπηρέτηση της προσπάθειας να συνεισφέρουμε με αυτή την αναθεώρηση υπέρ της απόφασης που υιοθετήθηκε από το Συμβουλίο των Υπουργών. Είναι ένα πρώτο σαφές συμπέρασμα. Η υπηρεσία αυτή είναι πλήρως λειτουργική και λειτουργεί σήμερα και πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αρετές και τις προσπάθειες της ΥΠΑ εκπροσώπου και των συνεργατών ιδιαίτερα του κυρίου Κρεμόν. Πρέπει μετά από αυτό να πούμε ότι πρέπει να διέπει μια λογική στη δράση σε ένα νομικό πλαίσιο τη δράση αυτού του, του μέσου με την απόφαση του Συμβουλίου δίνοντας τα αναγκαία μέσα και την αναγκαία φιλοδοξία ως πλαίσια. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε θαύματα, όμως θέλω να κάνω μια σύγκριση. Το προσωπικό δυναμικό και τα κονδύλια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρόμοια με εκείνα ενός κράτους μέλους όπως της Δανίας. Τούτου λεχθέντος μπορούν όλα βέβαια να βελτιωθούν και στο συντονισμό και στην εξωτερική δράση μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ενισχύοντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ΥΠΑ εκπροσώπου μέσω πολιτικών οργάνων, δίνοντας δυνατότητα στα Υπουργεία των κρατών μελών να συνδράμουν την ΥΠΑ εκπρόσωπο και να αναζητηθούν συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ε, κυβερνήσεων και διοικήσεων. Ένα καλό παράδειγμα η δράση της Ισπανίας στην Ιεμένη όσον αφορά την προξενική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Υπάρχει ένα θεμελιώδες ε, ε, στοιχείο, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό αυτών των διπλωματών ανακυκλώνοντάς τους και δίνοντας κίνητρα επίσης και στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινητοποιηθούμε με πολιτική βούληση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά και να ομιλεί με μία ενιαία φωνή και να έχουμε μία εξωτερική πολιτική που θα είναι πιο αποτελεσματική αποτελεσματική, πιο συνεκτική και πιο ευδιάκριτη. Και τα κράτη-μέλη για να αποφεύγουν μη ευκτές καταστάσεις, όπως είδαμε σε σχέση με τη συζήτηση για τη Συρία, να κατανοήσουν ότι πρέπει να αναζητήσουν τα προτερήματα στο κοινό συμφέρον που πρέπει να εξυπηρετείται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα. Κυρία Γκόμες τώρα, εξ των Σοσιαλδημοκρατών παρακαλώ να δημιουργήσουμε ένα ε, νέο όργανο ποτέ δεν είναι εύκολο έργο και γι' αυτό πρέπει να συγχαρούμε την κυρία Άστον και τον πρέσβη που πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αρετές και τα, και τα επιτεύγματά τους. Και για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, κάνουμε τα πρώτα βήματα προς μια πολιτική εξωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεκτική και αποτελεσματική. Χρειάζεται όραμα και φιλοδοξία ώστε η υπηρεσία αυτή να εξυπηρετεί μια κοινή πολιτική που θα αντανακλά ευρωπαϊκές αξίες και θα προασπίζεται και θα προαγάγει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκόσμια και εδώ δεν θα πρέπει να ε, υστερήσουμε από το να το αναφέρουμε αυτό και να το τονίσουμε. Είπατε εκπρόσωπος πρέπει να αναλάβει τον συντονισμό μεταξύ όλων των πολιτικών και μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επίπτωση στην εξωτερική δράση. Ασφάλεια, ανάπτυξη, εμπόριο, ενέργεια και όλα τα λοιπά. Ο θεσμικός χαρακτήρας απορρέει από τη διπλή ιδιότητα που έχει η ύπατος εκπρόσωπος και ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η διάφορη επίτροποι πρέπει να δεχθούν τον ηγετικό ρόλο που έχετε κυρία Άστον. Και εσείς πρέπει να είσαστε ηγέτης κυρία Άστον. Να χρησιμοποιείτε και να πιέζετε τους επιτρόπους αλλά και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επίσης. Χρειάζεται, πρέπει εδώ να επενδύσουμε στην κοινή πολιτική εξωτερική, ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Να διασφαλίσουμε ότι σε μια περίοδο κρίσης οικονομική να μην χάσουμε το δυναμικό μας και τις δυνατότητες μας. Θα πρέπει να εξορθολογήσουμε την χρήση των, του δυναμικού και των πόρων μα, ώστε να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι δράσει μα υπέρ τη ασφάλεια, συνολικά και σφαιρικά. Επίση, κατευθυντήριε γραμμέ σε όλε τι δράσει μα πρέπει να είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου, η προαγωγή τη ειρήνης και τη Δημοκρατία, παγκόσμια. Έχουμε ειδικό εντεταλμένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου τώρα. Πρέπει να προαγάγουμε αυτό και να δώσουμε ευδιάκριτο χαρακτήρα δίνοντα δυνατότητε, όπω απαιτεί αυτό το αξίωμα. Πρέπει ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, με στρατηγικούς εταίρους όπως με τη ΣΥΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και τη Βραζιλία, αυτά τα πλαίσια να είναι διαφανή και αποτελεσματικά όσον αφορά τους στόχους και τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων θα λάβει τον λόγο για δύο λεπτά επίση η κυρία Νέιτσα Οίτενμπρουκ παρακαλώ. Κυρία Πατή, εκπρόσωπε, με τις συνθήκες τη Αβώνα η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική άμεσης Ευρώπης ε, έχει ενοικηλικιωθεί ούτως υπήν και βάζει τα θεμέλια για πραγματικά μια κοινή διπλωματική ευρωπαϊκή υπηρεσία. Βέβαια δεν μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε διπλωματία, διότι μόνο τα κράτη-μέλη έχουν διπλωματία και διπλωματική υπηρεσία. Αποκαλείται λοιπόν υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν πρεσβείες Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά αντιπροσωπείες και οι επικεφαλείς τους δεν μπορούν να έχουν τον τίτλο πρεσβευτών είναι επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Για μην πνιγεί και ο Λόρδος Ντάτμουρ θα μου το πω αυτό. Λοιπόν, αποκαλύπτει αυτό τις ανησυχίες ε, των Υπουργείων Εξωτερικών των κρατών μελών και αρχικούς δισταγμούς που είχαν να συνεργαστούν με αυτή την πολύ νέα, το νέο δημιούργημα. Η απλή ύπαρξη λοιπόν μια εύρυθμα λειτουργούσα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερικής δράσης λιγότερο από τρία χρόνια από όταν άρχισε να υπάρχει, είναι θετικότατο στοιχείο αυτό κάθε αυτό. Και ένα θαυματάκι θα έλεγα και θα πρέπει να χαρούμε γι' αυτό. Βεβαίως υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων ο συνδυασμό τριών ιδιωτήτων, ε, είπα εκπροσώπου, Προέδρου της, του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών και Αντιπροέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που απαιτεί υπεράνθρωπη δύναμη και πανταχού παρουσία. Ξέρω ότι έχετε μεγάλη αντοχή, κυρία μου, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχουν περιθώρια για έναν ή, ή περισσότερους βοηθούς που θα μπορούσαν και πολιτικά να εκπροσωπούν τα, το λειτουργήμα του δυσύπατη εκπροσώπου. Χρειάζεται ευελιξία ούτως ώστε να γίνεται ιδέωσα προσαρμογή στις καταστάσεις που αλλάζουν γρήγορα και χρειάζεται να αποφευθεί αλληλεπικάλυψη και να μην υπάρχουν και συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε. Τώρα για δύο λεπτά στην παρέμβαση θα έχει την δυνατότητα να παρέμβει εξ ονόματος των Πρασίνων η κυρία Μπραντνερ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Άστον. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πράγματι πετύχατε πολλά την τελευταία τριετία και σας αξίζουν έπαινοι γι' αυτό. Συμφωνώ ότι μπορούμε πάντα να καταφέρουμε καλύτερα και θα πρέπει την αναθεώρηση αυτή να τη χρησιμοποιήσουμε σαν σοβαρή άσκηση και όχι άσκηση επί χάρτου. Επί της ουσίας, ε, να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία, ένας από τους βασικούς στόχους ε, της υπηρεσίας και που προβάλλατε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ένα από του καλύτερου φορεί όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων, τη διαχείριση των κρίσεων, την ανταπόκριση στα προβλήματα και λύση. Στη Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο τι είπατε. Μιανμάρ, Βιρμανία, Ιεμένη, γίνονται συγκρούσεις, δεν ακούμε πολλά για αυτά, αλλά έκανε πολύ καλή δουλειά η υπηρεσία. Πιστεύω ότι για να είμαστε ακόμα καλύτεροι θα πρέπει να πάρετε το ρόλο σας σαν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα πιο στα σοβαρά και δεύτερον, πιστεύω ότι πράγματι θα πρέπει οι αμυντικές δομές να ε, ολοκληρωθούν καλύτερα. Το συζητήσαμε με τον κύριο Ποπόσκι και μας είπε ε, εγώ ε, έχω τη δομή την οποία συμφωνήσαμε εδώ και τρία χρόνια και θα βάζω τη δουλειά που έκανε. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν είναι δομή, είναι άτομο. Είπε είμαι δομή. Του λείπει υποστηρικτική δομή. Λοιπόν ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί η κατάλληλη δομή το συζητήσαμε αυτό πριν από τρία χρόνια και εξακολουθώ να είμαι πεπισμένη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει να ανταποκρίνεται καλύτερη η Ευρωπαϊκή Ένωση στις, να αντιμετώπιση των κρίσεων και να επιβάλλει μακροπρόθεσμη ειρήνη. Και κάτι άλλο που αναφέρατε και χαίρομαι γι' αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολλή επικάλυψη Πολλά γίνονται σε υψηλό επίπεδο, πολύ λίγοι υπάρχουν επιτόπου και δεν υπάρχουν σαφεί διαχωριστικέ γραμμέ όσον αφορά το οποίο δίνει τι εντολέ και χαίρομαι που το είπατε ότι θα το θέσετε το θέμα αυτό στα πλαίσια του προπολογισμού του 2014. Αναφερθήκατε ισορροπία των δύο φύλων και υποσχεθήκατε ένα σχέδιο δράση που θα ασχολείται με τα θετικά εμπόδια για να επιτευχθεί ο στόχο. Υπάρχουν πολλά θετικά εμπόδια για τι γυναίκε όσον αφορά το διπλωματικό σώμα και θα ήταν καλό να μπορούσατε να δώσετε συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια στα πλαίσια τη αναθεωρήσεω. Τέλος, εσείς είστε ένα άτομο και έχετε τρεις ιδιότητες. Παρακαλώ προτείνετε και βοηθούς να μην πρέπει να κατηγορούμε ε, να σας κατηγορούμε ότι δεν είσαστε κάπου ε, γιατί πρέπει να είσαστε σε δύο-τρει άλλε συνεδριάσεις ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Ευχαριστούμε εξ ονόματος των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Για δύο λεπτά ο Δόκτωρ Τάνο. Πρόεδρε, στην αρχή εγώ ήμουν πολύ σταθερικό όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερική δράση που βεβαίω ε, μπορούσε να έχει μεγάλη εξουσία που θα έπαιρνε από τι εθνικέ κυβερνήσει. Όμω κάπω είμαι πιο μετριοπαθή. Και τώρα είδαμε ότι ανεπτύχθηκε όλος φορέας μέσω της καθιάς τον δίνει προστιθέμενη αξία όσον αφορά τι συνένεση που χρειάζεται σε εξωτερική πολιτική, πολιτική άμυνα, ανθρώπινα δικαιώματα και όλα κάτι τη της Ευρωπαϊκής που μιλάμε με μια φωνή και όπου δεν υπάρχει σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ. Τέτοια παραδείγματα είχαμε στην οργάνωση κυρώσεων κατά του Ιράν και του ποινικού προγράμματο, έξω και δουλειά που έγινε τη UNAF Αταλάντα και μειώθηκε δραματικά η πειρατεία στις ακτές της Ομαλίας, η δουλειά που κάνει η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο Ομαλή, τη Βυρμανία και πρόσφατα έγινε έγιναν πολλά επιτεύγματα στη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Και είπα ότι εκπρόσωπο ε, πρέπει να τύχει συγχαρητηρίων εκ μέρου μου. Επιτυχίε είναι αυτέ και ακριβώ αυτό θέλουμε αυτή την υπηρεσία. Θέλουμε οικονομία κλίμακα μέσω τη οργανώσεω που κάνει μια χρήσιμη δουλειά με καθορισμένε παραμέτρου. Γι' αυτό είναι λυπηρό που αυτή η έκθεση προσπαθεί να διευρύνει την εντολή τη υπηρεσία πέρα από αυτού τι αρχικέ προδιαγραφέ και αυτό ε, ουσιαστικά αποσπά διάφορε εξουσίε. Δεν μπορούμε να διεκτούμε ε, δεν θα μπορεί να έχουμε battle groups αναπτύσσονται σε δυνάμεις ταχείας αντίδρασης διότι θα είναι βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα που θα φέρουν το φόρτο εργασία και λέει η έκθεση ότι θα πρέπει σε θέματα ΚΕΠΑ να μην υπάρχει πλέον ομοφοφιγωνία και ήδη Γάλλοι, τα γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα θα μπορούν να πηγαίνουν στη μάχη με ειδική πλειοψηφία χωρί να συμφωνούν οι εθνικέ κυβερνήσει. Οι πολιτικοί σου τη πολιτική είναι ροχοκαλιά τη εθνική κυριαρχία και τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικέ προτεραιότητε, προπολογισμού και γεωπολιτικά συμφέροντα και στρατηγικά συμφέροντα. Και είναι απαράδεκτο να υποχρεώσουμε εμεί συγκεκριμένη χώρα ε, να παίρνει αποφάσει που είναι πάρα πολύ δαπανηρέ και επικίνδυνε κατά των εθνικών συμφερόντων. Το ECR απορρίπτει τη μείωση τη συμμετοχή των 100 μελών στο Συμβούλιο. Η, εναλλακτική εναλλαγή τη Προεδρία στο Συμβούλιο είναι ένα βασικό στοιχείο και αν σταματήσει αυτό ο ρόλο, αυτό θα προσθέσει πολεμοφόδια σε εκείνου που λένε ότι υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας και ελέγχου εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των δομών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και τέλος, η κληρονομιά της Relax θα πρέπει να εξεταστεί, γιατί δεν υπάρχει αντιπροσωπεία στο Παναμά της Relax, αλλά υπάρχει μεγάλη στους Μπαρμπέιντος. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Έχουμε μπλε κάρτα τώρα. Αλέξανδρε, Αλεξάνδρε, θα σου δώσω τον λόγο δεν δίνω τον λόγο για μπλε κάρτα σε εκείνους που θα παρέμβουν στη συνέχεια. Εντάξει, λοιπόν, διαφορετικά δεν θα τελειώσουμε έγκαιρα. Και πρέπει να τελειώσουμε έγκαιρα στις παρεμβάσεις. Γιατί διαφορετικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, τα επιχειρήματα ή ερωτήσεις έναντι του κυρίου Τάνοκ. Εντάξει, λοιπόν, για 1,5 λεπτό στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος Ντάρτμουθ, ο κόμις του Ντάρτμουθ. Παρακαλώ. Ε, η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Ενώσεω είναι η εξωτερική υπηρεσία υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και αυτή η υπηρεσία βασίζεται επί τη υποθέσεω ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ των 27 κρατών μελών. Αυτό όμω είναι σφαλμένο. Στη Λιβύη μόνο 8 ευρωπαϊκέ χώρε συμμετείχαν σε επιχειρήσει, όχι 27. Και μία από αυτές τις χώρες δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα 27 κράτη-μέλη είναι, πώς να το πω, μια συμμαχία των απρόθυμων και καμιά φορά και είναι λιγότερο και από απρόθυμη Υπάρχει και αυτή σπατάλη, φοβερή σπατάλη όσον αφορά την εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το προσωπικό της υπηρεσίας πληρώνεται με πολύ ψηλούς μισθούς. Μέχρι 100 υπάλληλοι απολαμβάνουν αμοιβέ που είναι μεγαλύτερες από αυτές ε, του Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας. Το οικονομικό κλίμα είχε κάποια συνέπεια. Δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο κλείνει πρεσβείες ε, και προξενία. Παρ' όλα αυτά υποχρεωνόμεθα να συμβάλλουμε και συμβάλλουμε με μεγάλα ποσά στην εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτως ώστε να προωθήσουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν, και επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μας. Και όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία Εξωτερική Δράση αποδεικνύει ότι η συμμετοχή τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει στην πράξη την επιρροή μα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Για ένα λεπτό τώρα, εξ ονόματο Ενωτική Αριστερά, ο κύριο Βίλι Μάγερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, η ομάδα μα είχε πολλέ επιφυλάξει και συνεχίζει να τι έχει για τη δημιουργία αυτή τη υπηρεσία εξωτερική δράση, για τη δομή, για την εντολή και επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί όπω θα έπρεπε να ελέγχεται άμεσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Και γενικά η εξωτερική πολιτική οποιασδήποτε χώρα μέλου πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο φυσικά των εθνικών κοινοβουλίων. Δεν συμβαίνει εδώ αυτό και έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εδώ επικαλύπτονται υπηρεσίε ε, όσον αφορά την, πολιτική, την εξωτερική πολιτική των κρατών μελών και τη ίδια εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια δομή που θα έπρεπε να έχει ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επ' αυτής για να ελέγχει. Και πόρο απέχουμε, κυρίε και κύριοι, από μια εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας ε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Είναι μια αλήθεια αυτή και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια εξωτερική υπηρεσία που θα υποστηρίζει αυτή την πολιτική, μια πολιτική κοινή ασφάλειας για όλους ε, που ελπίζουμε μακάρι, μακάρι να ήταν μια τέτοια εξωτερική πολιτική που θα βασιζόταν στον αφοπλισμό, στην αποστρατιωτικοποίηση και την επίλυση και αντιμετώπιση σειράξεων και προβλημάτων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, έτσι ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στον των αγοριτών εξ ονομάτων των ομάδων. Περνάμε τώρα στους συναδέλφους που ατομικά θα παρέμβουν. Πρώτα απ' όλα θα παρέμβει για 1,5 λεπτό ο κύριος Αντιπρόεδρος Προτασιέβιτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα, Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπο ε, να πω ότι ξεκινώ λέγοντα ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση που ξεκίνησε από μηδενικού σημείου πριν από 2,5 χρόνια απέδειξε ότι είναι χρήσιμη και αποτελεσματική. Και για να δικαιολογήσω αυτόν τον ισχυρισμό μου μπορώ να σα πω δύο λόγια για την κατάσταση που αφορά τη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο και το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου από πλευρά του Ιράν και το πρόβλημα των, της πειρατείας στη Σομαλία. Και ακριβώς ε, ως αντιπρόεδρος που αφορά, που ενδιαφέρεται για την ανατολική ε, εταιρική και γειτονική σχέση, ικανοποιούμε για το ότι η εταιρική ε, σχέση γειτονίας με τα ανατολικά κράτη είναι και αυτή ο συνιστός παρούσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, σε σχέση με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες ανατολικής γειτονίας, πρέπει πάλι να κρίνουμε τα πράγματα με θετικό τρόπο. Ωστόσο εδώ θα ήθελα να σας ζητήσω να ενισχύσετε, να ενδυναμώσετε τον ρόλο και την θέση των αρχηγών αντιπροσωπιών δίνοντας συγκεκριμένο έργο σε ε, χαμηλότερο επίπεδο ώστε οι ίδιοι αρχηγοί των ε, αντιπροσωπιών να μπορούν να ασχοληθούν με ανώτερα ε, θέματα υψηλότερης, μεγαλύτερης εμβέλειας. Θέλω επίσης να αναφέρω την άποψη της Amnesty International που λέει για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λιγότερο αποτελεσματική σήμερα από ό,τι πριν ε, τη, δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η κυρία Γιάκον Σάρη παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε στον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα και που ανακατανέμονται εξουσίες και αρμοδιότητες είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ομιλεί με μία ενωμένη ενιαία φωνή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική υπόθεση να είναι πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εργάστηκε ε, με ιδιαίτερα έντονο τρόπο η Λέδη Άστον για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Υπάρχουν όμως ε, και θέματα τα οποία οδηγούν στο να είσαστε υπομοιρία ομοιρία αυτής της τεράστιας γραφειοκρατικής δομής και έτσι δεν μπορέσατε να υλοποιήσετε όλους τους στόχους σας. Πρέπει να πάψει αυτό το γραφειοκρατικό βάρος, αυτή η γραφειοκρατική επιβάρηση. Πρέπει να σταματήσουν οι διπλοεπικαλύψεις. Πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι και τα κράτη-μέλη για τον, την πιο αποτελεσματική δράση. Ένα στοιχείο επί του οποίου θα ήθελα να τοποθετηθώ είναι ότι πρέπει να φέρουμε κάνουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση πιο κοντά στου πολίτε μα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν βελτιώσουμε την προξενική μα δράση υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι Αυστριακού και Φιλανδέζα που απήχθηξαν στην Ιεμένη δεν, είναι, δεν γνωρίζω αν ήταν πραγματικά υπόθεση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση ή των κρατών μελών για την απελευθέρωσή του. Θέλω να σα ευχαριστήσω όμω για τη δράση σα και τα θετικά αποτελέσματα αποτελέσματα. Για 1,5 λεπτό τώρα ο κύριο Λάμστορφ. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πριν από τρία χρόνια η Φρανσίσκα Μπράγνο και εγώ δημιουργήσαμε ένα θεσμό που είναι, αποκαλείται φίλοι τη Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Εξωτερική δράση, ώστε να μπορούν να συνέρχονται διπλωμάτε και αρμόδιοι για την ε, εξέταση των αναγκαίων δομών. Κάποια από τα πράγματα που εξετάσαμε έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη όσον αφορά την εκπροσώπηση. Είχαμε είχαμε υποβάλει προτάσεις ε, για τους αρμόδιους που είχαν τότε αναλάβει τα πράγματα είναι ε, κάτι το οποίο σε σχέση με τη δράση της ΥΠΑ εκπροσώπου είναι πολύ δύσκολο να συγκεραστούν ε, τρία, τρεις διαφορετικοί στόχοι χωρίς να υπάρχει η αναγκαία συνδρομή και επικούρηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναφέραμε. Το δεύτερο, κάτι το οποίο συζητήσαμε είναι μια ευρύτερη δομή ηγεσία αντί να υπάρχει ένας παντοδύναμος γενικός γραμματέας να υπάρχει μια μεγαλύτερη διάχυση. Δεν θέλαμε να υπάρχει κάποια θεά εξουσία ε, που θα βρίσκεται στα παρασκήνια. Θα θέλαμε να υπάρχει η δυνατότητα να αντλείτε τις περισσότερες πληροφορίες ε, για να είσαστε πιο αποτελεσματικοί και αυτή η αρχή νομίζω είναι, εξακολουθεί να έχει την αξία της. Το τελευταίο που ανέφερε ο συνάδελφος ε, ε κύριος Κόμις του ειναι είναι ότι κράτη-μέλη κλείνουν τις πρεσβείες τους και προξενία τους πολλές φορές και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα πρέπει να μπορεί να Εκπροσωπείται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την υπηρεσία εξωτερική δράση όπω πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Αλέξανδρε για την κατανόησή σου και για την ε, προσαρμογή σου στι ανάγκε μα ε, ω φίλο και συνάδελφο. Για 1,5 λεπτό κυρία Λούνατσεκ παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Άστον, κυρίες και κύριοι, και από πλευράς μου θερμά συγχαρητήρια προς την κυρία Άστον για την ομάδα σας και αυτά τα οποία καταφέρατε αυτούς τους τελευταίους μήνες και είναι επιτέγματα. Δεν ήταν καθόλου εύκολη δουλειά. Σας αναγνωρίζουμε τα θετικά και σας επενούμε. Διότι πού αλλού γίνεται να δημιουργείται από μια επιχείρηση μια ολόκληρη δομή και να προσδιορίζονται οι ανώτατοι αξιωματούχοι και μετά να δημιουργείται η κατώτερη δομή, περαιτέρω προς τα κάτω διάρθρωση. Σας ε, αξίζουν συγχαρητήρια και έπαινοι. Πραγματικά υπεράνθρωπος θένος και δυνατότητες απαιτούνται για να ε, καταφέρει κανείς να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Εκφράζω τη θλίψη μου το ότι δεν μπορούν να αποκαλούν πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι, εκπροσω... οι αντιπροσωπείες μας στο εξωτερικό αλλά είναι μόνο γραφεία εκπροσώπησης. Καταφέρατε επίσης στη Σερβία τους Σέρβους και τους να τους οδηγήσετε σε στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Αυτό είναι ιστορικό επίτευγμα και θα το καταγράψει και θα το αναφέρει και η ιστορία στις δέλτους της μελλοντικά. Εδώ υπάρχει και το δυναμικό της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Δύο από αυτά τα στοιχεία θα αναφέρω που δεν είναι ε, στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης αλλά αφορούν τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της ομοφωνίας στο Συμβούλιο και τη τάση, την τάση των μεγαλύτερων κρατών που δεν επιθυμούν ουσιαστικά η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να έχει κέριο ρόλο και σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική. Δεν φταίτε όμως εσείς γι' αυτό, δεν είσαστε εσείς ένοχος, άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την τάξη πραγμάτων. Τώρα για τις δομές, για εκπροσώπους σας στο μέλλον ή για τον ή την διάδοχό σας στο μέλλον που θα πρέπει να αναλάβετε δράση. Βλέπω τον αγώνα που δίνετε γυναίκες να ανέλθουν, να αναρριθούν στα ανώτατα κλιμάκια στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και είναι δουλειά όμως και των κρατών μελών να διορίσουν γυναίκες ώστε να εκπροσωπούν γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Έχεις ξεπεράσει το χρόνο σου. Για ένα λεπτό ο κύριος Κόμαλ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Παρακολουθώ το έργο της ε, υπηρεσίας στις χώρες που επισκέπτομαι συχνά, Ουκρανία, Μολδαβία, Λευκορωσία. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλες χώρες. αλλά αυτές αποτελούν πετυχημένα παραδείγματα. Η υπηρεσία είναι πλέον κομμάτι του ευρωπαϊκού τοπίου και θα ήθελα να θεωρήσω την υπηρεσία σαν εταίρος στην κοινή Ευρώπη του μέλλοντος. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την υπηρεσία τεχνητά. Ας ε, κάνουμε μια προσπάθεια μετριοπαθή. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το πνεύμα συνεργασίας ε, και η ενωμένη δράση θα βοηθήσει Μιλάτε πάρα πολύ ωραία για τα δικαιώματα των γυναικών. Γιατί να μιλάμε και για τα δικαιώματα των χριστιανών. Διώκονται σε πάρα πολλές περιοχές. Χρειάζονται τη φωνή σας, την παρέμβασή σας, ε, ε, Επίτροπε. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη ισορροπία, διότι η Πολωνία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε στατιστικό, στατιστική άποψη. Για να υπάρξει επιτυχία και στη χώρα αυτή πρέπει να τηρήσετε την ισορροπία. Σας ευχαριστούμε κύριε Για ένα λεπτό πάλι ο κύριος Φανχέκε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Λυπούμε που θα πρέπει να διαφωνήσω σε σχέση με αυτή την συνένεση που εκφράζεται στην Ολομέλεια. Πρόκειται για μια ειδική μελέτη περίπτωσης ε, πώς δεν θα έπρεπε να δράσουμε ιδιαίτερα με πράγματα τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ε, άρδιν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα ε, ήμουν σε θέση να μπορέσω να υποστηρίξω το αίτημα υπέρ των βελτιώσεων. Όμως όχι, να μην θεραπεύσουμε μόνο τα συμπτώματα αλλά και τα αίτια. Αλλά ακόμα και αν πραγματικά ε, θα αποχωρήσει η κυρία Άστον, ακόμα και αν αντιμετωπίσουμε τον υπερβολικό αριθμό Ευρωπαίων διπλωματών που πληρώνονται υπερβολικούς μισθούς, τα θέματα αυτά παραμένουν ως έχουν. Δεν είναι φεντεραλιστικής δομής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε εκφράζει μία ενιαία ε, εξωτερική πολιτική ή μία ενιαία διπλωματία. Μπορεί να εκφράζει κανείς τη θλίψη του για αυτή την κατάσταση, όμως είναι δεδομένη και εφόσον είναι δεδομένη δεν έχουμε το δικαίωμα να ρίχνουμε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ένα εγχείρημα το οποίο είναι περιττό και δεν ωφελεί σε τίποτα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό θα παρέμβει τώρα ο κύριο Ντανζόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε, είπατε εκπρόσωπο η υπηρεσία εξωτερική δράση και η θέση που κατέχετε σήμερα είναι ε, αποτελέσματα θετικά τη συνθήκη τη Λισαβόνα παρά τι ατέλειε, παρά τι αναγκαίε προσαρμογέ και τι κριτικέ που ακούγονται συχνά, α μην ξεχνάμε ότι όταν ζητάμε από του συμπολίτε μα, ποια είναι, είναι το οποίου θα ήθελα να βλέπουν να παίζει συλλογικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο ενεργό ρόλο, η διπλωματία και η ασφάλεια και η άμυνα αποτελούν τι προτεραιότητε που μα αναφέρουν. Είναι λοιπόν θετικό που βλέπουμε αυτή την εξέλιξη και σε βέβαια σε τρία χρόνια δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό διπλωματικό σώμα, μια κοινή ε, διπλωματία. μετά από αυτά που μας είπαν η συνέκτασή τους οι κύριοι Μπρόκ και Γκουαλτιέρη θέλω να επιμείνω ειδικότερα σε αυτό που αφορά τις πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την ιδιότητά μου συνάντησα όλους τους αρχηγούς αποστολών, επισκέφθηκα όλες τις αποστολές, διαπιστώνω δυστυχώς πάρα πολύ συχνά το ίδιο πράγμα. Προγραμματισμός, σχεδιασμός που είναι ε, ανεπαρκής, ένα συντονισμός που είναι επίσης ανεπαρκής, μια ευελιξία που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Πρέπει να βελτιώσουμε οπωσδήποτε την κατάσταση διότι από αυτό εξαρτάται η αξιοπιστία και η προβολή μας. Κυρία είπατε εκπρόσωπο, θα είναι επιμείνω στο ρόλο που έχετε ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Τα γρανάζια της Επιτροπής και η χρηματοδότηση της Επιτροπής πρέπει να χρησιμοποιούν με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο υπέρ των εξωτερικών μας αποστολών. Ευχαριστούμε κύριε. Σας ευχαριστούμε κύριε Για ένα λεπτό η κυρία Μαρία Μουνίτ Ντεουρκίθα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω σε σχέση με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα θετικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> να αποφύγουμε διπλοεπικαλύψει ε, με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, για παράδειγμα, και να γίνει πιο ελαστικό ο ρόλο ε, τη ΥΠΑ εκπροσώπου, ώστε να μην έχει αυτή την ε, δίσκαμπτα διτή ιδιότητά τη. Και από την άλλη πλευρά, σε σχέση με τα θετικά στοιχεία, πρέπει να είμαστε και πιο φιλόδοξη σε σχέση με την εξωτερική δράση, δίνοντας ε, επιλογή και προτεραιότητα σε σχέση με τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να κλείνουν τις, ε, κλείνουν τις πρεσβείες τους ε, προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν όλοι ότι είναι μια ωφέλιμη, χρήσιμη υπηρεσία που χωρίς να μειώνονται τα δικαιώματα υπέρ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες μπορούν να εκπροσωπηθούν τα συμφέροντά τους από την εξωτερική υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Επίσης να δούμε και την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στην εκπροσώπηση των γυναικών στους υπαλλήλους. Μηδενικό επίπεδο από το, ε, το ΑΔ16 έως χαμηλότατα ποσοστά στο ΑΔ13 και 70% στις βοηθούς που είναι όλες οι γραμματείς γυναίκες στη συντριπτική πλειοψηφία. Πρέπει εδώ λοιπόν τη δέσμευση που έχετε αναλάβει υπέρ της εκπροσώπησης των γυναικών και είναι και δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι γι' αυτό. Σε σχέση με το ΕΛΚΑ, σε σχέση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, λυπάμαι που απορρίφθηκε μια τροπολογία στην κοινοβουλευτική μας Επιτροπή που υπενθύμιζε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο υψηλότερο επίπεδο ποσοστώσεων υπέρ των γυναικών. Διακόπτεται η ομιλήτρια. Τώρα θα λάβει τον λόγο για ένα λεπτό επίση, η κυρία Γιάταν Μέκη. Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την έκθεση που προωθεί την υπηρεσία εξωτερικής δράσης διότι στηρίζεται σε γεωγραφική ισορροπία και αυτή η γεωγραφική ισορροπία είναι ιδιαίτερα σημαντική και σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται με ισότιμο και ισόρροπο τρόπο σε αυτή την υπηρεσία. Δυστυχώς σήμερα η κατάσταση είναι τέτοια που επικρατούν μόνο ορισμένοι στην υπηρεσία. 14% είναι Γάλλοι, ασφαλώς καλοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν εξαιρετικούς διπλωμάτες. Όπως είπε μόλις η Λέδη Άστον, 18% προέρχονται από 12 νέα κράτη-μέλη. Η άλλη όψη του νομίσματος ωστόσο είναι ότι από, το, μεταξύ, 15, 15 χώρες προσφέρουν, προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό ε, των μελών της υπηρεσίας. Πρέπει λοιπόν να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ στη συνέχεια κύριος Πιοτρόφσκι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ στην ε, εξέταση της λειτουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης mm. πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει γεωγραφική ισορροπία. Στην έκθεση, στο αντίστοιχο άρθρο, τονίζει το Ευρωκοινοβούλιο την ανάγκη να χρησιμοποιούνται όλες οι δράσεις και τα μέσα ώστε να διασφαλίζεται και να εισάγεται η γεωγραφική ισορροπία σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα αξιώματα. Ωστόσο, απουσιάζει αυτή η ισορροπία σήμερα. Διπλωμάτες από τα κράτη-μέλη και από την Πολωνία είναι ένα, ένας πολύ μικρός αριθμός ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, αν συγκρίνεται τον αριθμό τους με τους διπλωμάτες των εντός εισαγωγικών παλαιότερων χωρών. Η Πολωνία που είναι η μεγαλύτερη από τις καινούριες χώρες ε, από τις, στις αντιπροσωπείες δεν θα πρέπει να έχουμε τέσσερα τέτοια αξιώματα αλλά δώδεκα και, βρισκό, και δεν θα πρέπει να είμαστε στα χαμηλότερα αξιώματα αλλά και σε υψηλότερα. Από 3.000 θέσεις ε, βλέπουμε ένα ποσοστό 3% συνολικά. Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν η γεωγραφική ισορροπία θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα σοβαρά με τη θέσμιση εθνικών ποσοστώσεων. Ευχαριστώ συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Πρέντα παρακαλώ. Πρόεδρε, Είμαι ευτυχής επειδή οι συστάσεις Μπρόκ και Κουαλκέρι υπογραμμίζουν ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι μια νέα υπηρεσία και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα λειτουργεί ε, τέλεια 100% τους τα πρώτα δύο, τρία, τα δύο-τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. Ορισμένοι συνάδελφοι υπήρξαν ιδιαίτερα σκληροί απέναντι στην κυρία Άστον λόγω των ε, περιορισμών που αντιμετωπίζει στα πλαίσια αυτής της διαδικασία. Η λέξη κλειδί θα έπρεπε να είναι εδώ ευελιξία. Ευελιξία σε ό,τι αφορά την ανακατανομή των πόρων και του προσωπικού τη στιγμή της αλλαγής των πολιτικών προτεραιοτήτων όπως το ε, ε, ε, έδειξαν και χώρες ταχεία παρέμβαση και μεγαλύτερη ευελιξία για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας ε, όπως διαπιστώσαμε ε, με την περίπτωση της κρίσης στο Μαλί. Θα ήθελα παράλληλα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι έστω και αν η υπηρεσία δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την εθνική διπλωματία, αυτή η υπηρεσία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο στο οποίο σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν περικοπές δημοσιονομικές για οποιαδήποτε διπλωματική εκπροσώπηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Για ένα λεπτό στη συνέχεια ο κύριος Κράισαλντόρφερ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάνουμε μια ενδιάμεση αξιολόγηση και επανεξετάζουμε ποιες δομές ήταν οι πιο θετικές για αυτή την υπηρεσία και πού υπάρχει δυναμικό για βελτιώσεις. Ένα πράγμα σε σχέση με τις κρίσεις ε, που αντιμετωπίσαμε πέρσι είναι σαφές. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική ηγεσία από πλευρά της ΥΠΑ της εκπροσώπου ώστε να είμαστε σε αποτελεσματικό επίπεδο στην εξωτερική μας πολιτική. Αξιότιμη κυρία Άστον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλύτερα αυτό το δυναμικό και ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και σε σχέση και με τα μέλη της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θα σας υποστηρίξουμε στις πρωτοβουλίε σας σε όλα αυτά τα διαβήματα και παράλληλα προς μια πιο ενισχυμένη ηγετική ε, ε, δραστηριοποίηση θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είναι αποφασιστική σημασία το, ο τομέας της ε, πολιτικής γειτονίας να παραμείνει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να έχουμε την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ' αυτής. Δεν μπορεί να γίνεται σε διακυβερνητικό επίπεδο. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι για το έργο που επιτελέσατε. Εξαιρετικούς συνεργάτες έχετε, γυναίκες και άνδρες. Και θέλω ιδιαίτερα τον συνάδελφο εξεβονίμων σας να αναφέρω τον κύριο Ρέμον που είναι εξαιρετικό στο έργο που έχει επιτελέσει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Βόλφ. Για 1,5 λεπτό κυρία Γιαννάκου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι αλήθεια ότι η δημιουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προσέφερε πάρα πολλά θετικά μέχρι στιγμής και θέλω να συγχαρώ την κυρία Άστον για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει γιατί η υπόθεση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη. όμως παρακολουθώντας το πώς έχει λειτουργήσει η υπηρεσία νομίζω ότι πρέπει να δεχθεί κανείς ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να αλλάξουν όπως προτείνει το κοινοβούλιο. καταρχήν η ιεραρχική δομή πρέπει να τύχει καλύτερης εφαρμογής. φαίνεται πως υπάρχει μια υπερφόρτωση από ανώτερους υπαλλήλους και φαίνεται πως πολλές φορές υπάρχει ένας ε, συγκερασμός των προσπαθειών όχι απόλυτα συντονισμένος μεταξύ της ευρωπαϊκής επιτροπής γενικά και της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. έχω την εντύπωση λοιπόν ότι μαζί με μια προσπάθεια να υπάρξουν περισσότερες γυναίκες οι οποίες εκπροσωπούνται δυστυχώς στην υπηρεσία αυτή ε, και με την εγκατάσταση ενός βασικού στρατηγίου στις βρυξέλλες και για την ασφάλεια και την άμυνα είτε για στρατιωτικές είτε μη στρατιωτικές δράσεις ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης της ένωσης θα έχει να επιδείξει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να αντιδράσει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και βεβαίως κύριε πρόεδρε επαναλαμβάνω ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει και τον αγώνα που γίνεται και βάσει αυτών των προσπαθειών ζητούμε να υπάρξουν ουσιαστικότερες αλλαγές τέτοιες που θα κάνουν την ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης να συντονιστεί καλύτερα και κυρίως να δείξει τα αποτελέσματα γιατί η ένωση πρέπει να αποκτήσει ένα brand name στο εξωτερικό που δεν το έχει ακόμα. είναι δυσανάλογα αυτά τα αποτελέσματα σε σχέση με τις ουσιαστικές προσπάθειες που υπάρχουν. εκεί λοιπόν χρειάζεται μια μεγαλύτερη προώθηση. ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό ο κύριος Κορτές Λάστρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπα το εκπρόσωπο κύριε Άστον για την εξαιρετική διπλωματική δουλειά που έχει επιτελέσει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Και να αναγνωρίσω επίση ότι είναι μια νέα υπηρεσία και λαμβάνοντα υπόψη και διάφορε πτυχέ τη λειτουργία τη. Ω μέλο τη Επιτροπή Ανάπτυξη, ε, περνώ το γεγονό ότι είπα ότι εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο στρέφεται ετήσια ε, στην ε, δική μα κοινοβουλευτική επιτροπή όσον αφορά τι δικέ μα αρμοδιότητε τη ανάπτυξη ενδιάμεση αξιολόγηση ελπίζω ότι θα αναλύονται αυτά τα πράγματα όπως πρέπει. Κυρίως μια βελτίωση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και των πολιτικών. Θέλω να δώσω ενθάρρυνση και να προτρέψω παρόλες τις ε, δυσκολίε, αρχικές δυσκολίες, να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός των πολιτικών μας στο εξωτερικό επίπεδο με τις πολιτικές ανάπτυξης, ώστε από κοινού να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην προαγωγή των θεμάτων ανάπτυξη. Και Επίσης θέλω να υπάρξει και μια ισορροπία και γεωγραφική και των κρατών μελών και των φίλων σε αυτήν την υπηρεσία. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό θα λάβει τον λόγο ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να είναι ένας ισχυρό πυλώνας της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Για αυτό το σκοπό Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερη χρήση των διαθεσίμων πόρων. Είναι μια νέα δομή, ε, εξακολουθεί να είναι νέα, είναι ένα εργοτάξιο κατά κάποια έννοια. Τα τελευταία χρόνια είδαμε επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, αλλά διαπιστώθηκαν και κάποιες ελλείψεις και αυτές θα πρέπει να καλυφθούν. Χρειαζόμαστε ισχυρό καλύτερη υπηρεσία, αποτελεσματικότερη υπηρεσία, χρειάζεται να ηγούνται στο πολιτικό προσκήνιο. εξωτερικέ σχέσεις και η πολιτική γειτονία είναι τομεί όπου η Ένωση μπορεί να δραματίσει πολύ βασικό ρόλο. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε με μια ισχυρή φωνή, φωνή που θα γίνεται σεβαστή. δεύτερον, αυτή η δομή της υπηρεσίας θα πρέπει να υποστηρίζει την εφαρμογή των εξωτερικών πολιτικών. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τις προσφερόμενες ε, δυνατότητες και να αποφύγουμε αλληλεπικάλυψη εργασιών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα πρέπει επίσης να βοηθούν τη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα χρειαζόμαστε μια διαφανή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη γνωμοδότησή του θα πρέπει να λαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο συχνά υπόψη όταν λαμβάνονται αποφάσεις. Διότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, βοηθά διαφάνειες δραστηριότητές σας και έτσι πλησιάζει η δραστηριότητά σας και τους πολίτες. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη δημογραφική ισορροπία στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και θα ήθελα να υπενθυμίσω Βαρόνι Άστον για τις δυνατότητες που έχουν και οι διπλωμάτες από την άκρα τη μέλη. ευχαριστούμε Έντουαρντ. Και τώρα για 1,5 λεπτό θα λάβει τον λόγο αντιπρόεδρος κύριος Οτμαρ Κάρας. Παρακαλώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι, αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους, τους πολίτες τι θέλουν και τι περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν κυρίως μια κοινή εξωτερική πολιτική. Μια σαφής αρμοδιότητα με σαφές πρόσωπο, ευδιάκριτο χαρακτήρα στην εξωτερική πολιτική από πλευρά της Ευρώπης. Αν δει κανείς τις εξελίξεις και τις ε, επιπτώσεις τη παγκοσμιοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> είναι πρέπει να γίνει να αποκτήσει ευδιάκριτο χαρακτήρα και να εκφράζεται ενιαία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν έχουμε μια αποτελεσματική υπηρεσία εξωτερικής δράσης, διπλωματική υπηρεσία. Πάρα πολλά πρέπει να γίνουν για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Βρισκόμαστε στην έναρξη, στην αρχή αυτών των βημάτων, αλλά δεν πρέπει να υπάρξουν ε, στρεβλές εξελίξεις με κατακαιρματισμό όσον αφορά αρμοδιότητες ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των κρατών μελών και της δράσης της εξωτερικής υπηρεσίας. Αυτό δημιουργεί αναποτελεσματικότητα και γι' αυτό ο κατακαιρματισμός αυτός πρέπει να καταργηθεί, να αρθεί. Εδώ σε ένα δοκίμιο της συναδέρφου Ingrid Gressler έχουμε και το οργανόγραμμα σε ανάλυση που δείχνει αυτό το οργανόγραμμα πόσο κατακαιρματισμένος είναι ο χαρακτήρας και δυσδιάκριτος ε, στις δράσεις. Ακούω από κάποιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ότι υπάρχουν και διαφορετικές περίοδοι διακοπών για τους υπαλλήλους. Διαφορετικά επίπεδα δράσης. Αυτά όλα πρέπει να καταργηθούν. Το Κοινοβούλιο θα είναι πάντα στο πλευρό όταν θα προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια αυθεντική υπηρεσία εξωτερικής δράσης και να καταργηθεί αυτός ο κατακαιρματισμός επιτέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Αντιπρόεδρε Κάρας. Ε, Κύριε Πέρετ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πετύχει πολλά μέχρι σήμερα, αλλά πολλά πρέπει να γίνουν και απομένει να γίνουν ακόμα. Γεωγραφική ισορροπία στα αξιώματα, σημαντική υπόθεση. Επίσης, ε, να υπάρξουν περισσότερα στελέχη και συνεργάτες από τα νέα κράτη-μέλη σε σχέση με τα παλαιότερα. Εδώ οι αρμοδιότητες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και οι ικανότητες πρέπει να είναι τα κυριότερα κριτήρια. Επιπλέον, πέρα από αυτά, θα πρέπει οι ηγετικές τα ηγετικά αξιώματα να έχουν και δεξιότητες και ικανότητες ξεχωριστές και σε σχέση με πρέσβεις έχουμε δει ότι δεν μπορούν πολλές φορές να επικοινωνήσουν, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία έχουν αποσταλεί. Για παράδειγμα, στην αντιπροσωπεία στη Μόσχα και με την προσπάθεια ανάληψης ε, επαφών. Δεν μπορούσαμε να έχουμε τέτοιες επαφές, δεν γινόταν να επιτευχθούν αυτές οι επαφές, διότι υπήρχε έλλειψη, απουσία επικοινωνίας και στο γλωσσικό επίπεδο και οι εκπρόσωποι των βαλτικών ε, κρατών, για παράδειγμα σε σχέση με τις αντιπροσωπίες ε, όσον αφορά τις χώρες της ε, ανατολικής γειτονίας ε, θα έπρεπε να μπορέσουν πραγματικά να προσληφθούν. Αυτό θα έδειχνε ότι θα είχαμε περάσει μια ολόκληρη καινούρια καμπή σε μια νέα πορεία. Και στο Τουρκμενιστάν η αντιπροσωπεία που είναι πολύ σημαντική αυτή η χώρα, όχι μόνο φυσικά λόγω των πόρων, φυσικών πόρων που έχει, αλλά και γεωπολιτικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Περισσότερα κονδύλια λοιπόν για προξενικές, ε, προξενικές και για τις μικρότερες χώρες είναι πολύ σημαντική υπόθεση. η, η, Αυτή η υπηρεσία είναι σημαντική για την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο που ενισχύεται παρόλη την οικονομική κατάσταση και τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζονται. Πιστεύω ότι η υπηρεσία λειτουργεί έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να εκφράζεται καλύτερα, να ακούγεται να, να, πιο πολύ, αλλά Πάρα πολλά πράγματα μπορούν ακόμα να βελτιωθούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλάει με μία φωνή, διότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος να αξιοποιήσει, να αξιοποιήσει και να προβάλλει τη θέση της στον κόσμο. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, που μου φαίνεται ιδιαίτερο σημαντικό για τη χώρα μου, τη Μάλτα. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, που κατέληξαν στην απόφαση της ίδρυσης της υπηρεσίας επιμείναμε στο γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος, ακόμα και τα πιο μικρά, θα πρέπει να εκπροσωπούνται σωστά. Εκτιμώ τις προσπάθειες που έχουν γίνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν προχωρήσαμε μέχρι το τέλος. Δεν ολοκληρώθηκε η προσπάθεια και θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές τα ερχόμενα χρόνια. Και χαιρετίζω το άρθρο 14 της σύσταση, όπου αναφέρεται ότι όλα τα μέτρα πρέπει να ληφθούν για να διορθωθούν οι γεωγραφικές ανισορροπίες σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης της υπηρεσίας διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε 7 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο και θα τον πάρουν αν όλοι τηρήσουν το χρόνο τους. Ε, πρώτα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, συνάδελφο Κόρχολα. Ευχαριστώ. Ανήκω στους ευρωβουλευτές που πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή εξωτερική πολιτική. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, ώστε να, φροντίζουμε, να μπορούμε να φροντίζουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως μας θύμισε μία συνάδελφος την δίωξη των ε, χριστιανών. Η υπηρεσία είναι σημαντική, η δομή της είναι σύνθετη, δεν μπορούμε να αναμένουμε θαύματα μετά από τρία χρόνια, αλλά η αντίδρασή μα στι κρίσεις υπήρξε αργή λόγω γραφειοκρατία. Υπάρχουν υπερβολικά πολλά επίπεδα λήψη αποφάσεων. Η Αραβική Άνοιξη και το Μαλί είναι, είναι δύο σημαντικά παραδείγματα. Ελπίζουμε όμως ότι μαθαίνει από τα λάθη της η υπηρεσία και βελτιώνει τι υπηρεσίε που παρέχει. Την περασμένη εβδομάδα η η εκπρόσωπος ε, για συνάντησε στην Τουρκία ε, την νεολαία. Πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη και το είχα ήδη τονίσει Θα ήθελα να επισημάνω κάτι ότι η πορεία προς την ευρωπαϊκή εξωτερική δράση είναι ακόμα πολύ μακρά και μεγάλη. Μία ερώτηση, γιατί αυτό το οργανόγραμμα εξακολουθεί να υφίσταται μια και η υπηρεσία εξακολουθεί και υφίσταται παρά αυτό το οργανόγραμμα και όχι λόγω του οργανογράμματος. Χαίρομαι για το ότι εδώ αναφέρατε το θέμα της αναδιάρθρωσης και προσδοκώ να δω τι θα γίνει. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τους ειδικού εντεταλμένους. Εκτός από τα έξοδα τα οποία τους καταβάλλονται υπάρχουν ε, κάποια αποτελέσματα. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι ειδικοί εντεταλμένοι. Ίσως θα έπρεπε να ενισχυθούν οι αντιπροσωπείες. Πρέπει να δώσουμε αγώνα για μια αποτελεσματική υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πληρώνουν 55.000 διπλωμάτες οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Είναι πολλαπλάσιο αυτό που, αυτόν που έχουν οι ΗΠΑ Ίσως θα ήταν πιο σκόπιμο να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα εξοικονομούσαν πολλά κονδύλια οι φορολογούμενοι με αυτόν τον τρόπο. Κυρία Πρόεδρε, οι ρυθμίσεις που προτείνει η έκθεση αποσκοπούν στην αναβάθμιση της υπηρεσίας ως πολιτικό στρατιωτικό μηχανισμό με μεγαλύτερη δύναμη πυρός για τις imperialistικές επεμβάσεις της ευρωπαϊκής ένωσης σε διεθνή κλίμακα να κάνουν την εξωτερική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης ακόμα πιο επιθετική πολιτική μόνιμων επεμβάσεων με ενίσχυση των στρατιωτικών χαρακτηριστικών της για διεξαγωγή εκτεταμένων πολεμικών επιχειρήσεων. η αναβάθμιση της υπηρεσίας προωθείται με μέτρα όπως καθιέρωση μόνιμου επιχειρησιακού στρατηγίου για επιχειρήσει κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, συμμετοχή των μάχημων μονάδων battle groups στι επεμβάσει Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτάχυνση των διαδικασιών χρηματοδότηση και λήψη αποφάσεων μέτρα για μόνιμη δομή διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων διαχείριση κρίσεων. με τη σύσταση πολιτικού συμβουλίου και μέτρα επίδραση πολιτικέ των κρατών μελών επιχειρείται να διασφαλιστεί ανεξέλεγκτη δράση τη υπηρεσία. το έτσι κι αλλιώ απαραγματοποίητο και υποκριτικό αίτημα για δήθεν ενημέρωση και έλεγχο του ευρωκοινοβουλίου στη δράση της υπηρεσίας μοναδικό σκοπό έχει να προσδώσει δημοκρατικοφανή δίθεν νομοποίηση στις στρατιωτικές επεμβάσεις της ευρωπαϊκής ένωσης και του νατο. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο συνάδελφος Μέλτσερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, Ποια αποστολή έχουν οι Ευρωπαίοι, κυρία Πρόεδρε, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν ένα κεντρικό μόρφωμα το οποίο θα δημιουργηθεί με κεντρικό χαρακτήρα και στους πολίτες των κρατών μελών, ας το πω έτσι, θα επιβάλλει δυναστικά τα κελεύσματά του ή θέλουν μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση με την αρχή της επικουρικότητας φιλελεύθερη, δημοκρατική και ισχυρή προς τα έξω που θα είναι σε θέση να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της, των πολιτών. Σίγουρα αυτό το δεύτερο θα επιλέγαμε και γι' αυτό θα πρέπει έτσι να διαμορφωθεί η κοινή εξωτερική μας πολιτική μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτό που έχουμε όμως σήμερα είναι μια αξιοπερίεργη διτή στρατηγική. Έχουμε τι παλαιές εντό εισαγωγικών μεγάλε δυνάμεις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Υπήρου που εξακολουθούν να ακολουθούν τις ξεχωριστές τους πολιτικές και θέλουμε να έχουμε μια εξωτερική πολιτική ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε όμως νάνοι. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει πρώτα να έχουμε μια σκόπιμη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή εξωτερική. Συνάδελφος Κρίσιπ. you, Madam Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οργάνωση της ε, υπηρεσίας αποφασίστηκε όταν ε, ε, λήφθη γιατί, για με σκοπό να υπάρχει μια εξορρόπηση δυνάμεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Διότι υπήρχαν, ε, υπήρχαν κάποιες ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από τα διάφορα θεσμικά όργανα. Επίσης έπρεπε να ληφθούν υπόψη γεγονότα όπως η Αραβική Άνοιξη έπρεπε να διοριστεί ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. Νομίζω λοιπόν ότι ε, ε, έχει αναπτυχθεί κατάλληλη συνεργασία με επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για την ανθρωπιστική βοήθεια και άλλα θέματα αλλά είναι σημαντικό και άλλοι επίτροποι να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία διότι η εξωτερική πολιτική πλέον δεν σημαίνει διαπραγμάτευση, δεν αφορά μόνο τη διαπραγμάτευση, αλλά και οικονομικά ζητήματα. Οι υπουργοί έχουν δυνατότητες να, προσφέρουν πολλά στην υπηρεσία. Το είπε αυτό η κυρία Άστον όταν αναφέρθηκε στην θετική επιρροή που άσκησαν οι διπλωμάτε των νέων κρατών μελών και την ευχαριστώ. Και τέλο, η συνάδελφος Σενκλέρ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλοί συνάδελφοι σήμερα ζήτησαν να ε, μιλάει με ενιαία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε εκπρεσβευτές αντιαρχηγούς αντιπροσωπιών αλλά αυτό απαιτεί κάποιο φεντεραλισμό, συνεπάγεται κάποιο φεντεραλισμό και δεν υπάρχει εντολή γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η υπηρεσία εξωτερική δράση θα αντιμετωπίσει προβλήματα και θα είναι δύσκολο για τη Βαρόνη Αύστον να εκπληρώσει τα καθήκοντά τη. Αισθάνομαι ότι ε, ευθύνεται εν μέρη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Όταν άσκησε πίεση για τη συνθήκη της Σαββόνας και είπε ότι έπρεπε να γίνουν σημαντικές αλλαγές και τώρα ζητάει περισσότερη ισχύ, περισσότερη δύναμη. Δεν μπορείτε να έχετε τα πάντα βαρώνει. Το να μιλάμε με μία φωνή σημαίνει ότι δίνουμε, ε, υπακούμε στην εντολή του λαού. Και αυτό που θα ήθελα να απαντήσετε απόψε είναι υπό ποια ιδιότητα, Βαρόνι Άστον, είσαστε στους ναι. τελικούς του Champions League φέτος. Um, Vice President... Και τώρα αντιπρόεδρος και ότι εκπρόσωπος έχει το λόγο. Ήμουνα στο τελικό κατόπιν προσκλήσεως της UEFA. να ευχαριστήσω όλου όσου πήραν το λόγο. Είπα και θεωρώ ότι θα ήταν ζωηρή συζήτηση και πράγματι αυτό ήταν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλιά σα. Είτε συμφωνείτε με αυτά που κάνουμε, είτε διαφωνείτε. Είναι σημαντικό το κοινοβούλιο, να, στο κοινοβούλιο να ακούγονται όλε οι φωνέ. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε κάποια από τα βασικά θέματα που εφήγησαν και να προσπαθήσω να απαντήσω. Βεβαίω θα επιστρέψουμε στο ζήτημα αυτό και στα ζητήματα αυτά δημοσιεύοντα την αναθεώρηση και θα ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά σε κάποια θέματα. Το πρώτο αφορά το πώς εργαζόμεθα και πώς συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Όπως είπα και στα αρχικά μου σχόλια, η Λισαβόνα άφησε το Συμβούλιο και τη διακυβερνητική ε, φύση και την ομοφωνία στα όσα κάνουμε, να επικρατούν για στα όσα κάνουμε. Θεωρώ ότι τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Υπουργοί Εξωτερικών, Υπουργοί Άμυνας, Υπουργοί Ανάπτυξης, θέλουν και είναι αποφασισμένοι να φτάσουν σε μια κοινή θέση. Όχι στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, αλλά στον ύψιστο κοινό παράγοντα. Ακόμα και αν αυτό είναι δύσκολο και όταν δεν υπάρχει συμφωνία, σας διαβεβαιώ ότι ο τρόπος με τον οποίο όλα και τα 27 κράτη-μέλη ε, συνεννοούνται, ε, είναι κάτι που οδηγεί σε μια συζήτηση πολύτιμη και αξιόλογη με επιδίωξη της λύσης. Αυτό ισχύει και για το 12ωρο που ξοδέψαμε για να συζητήσουμε τα θέματα για τη Συρία και το εμπάργκο. Άλλα μέλη έθεσαν κατά πόσο τα κοινοβούλια των κρατών μελών πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο. Κάθε προεδρία με την οποία συναντώμε βλέπω εκπροσώπους και από τα 27 κράτη-μέλη και από τα κοινοβούλια των 27 κρατών μελών έρχονται μαζεύονται και στην ενακτήρια συνεδρίαση έρχονται σε επαφή μαζί μου στη συνεδρίαση αυτή, στη Σύνοδο και συζητούμε επί μακρόν. Ίσως να μην αρκεί αυτό, αλλά σημαντικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς που κάνω. Όσον αφορά το πώς συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, πιο συγκεκριμένα, δόθηκε το παρά... Τι έγινε με, την... Ε, με τις απαγωγές στην Ιεμένη. Η Αυστρία και η Φιλανδία μας ευχαρίστησαν για τη δουλειά που κάναμε ε, σε επαφέ που είχαμε την κυβέρνηση, μίλησα με τον πρόεδρο και κάναμε προσπάθειε συντονισμού. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε θύμα ε, απαγωγής ε, υπήκο από κράτους μέλους. Οπουδήποτε και γίνει απαγωγή στον κόσμο, ζητάτε βοήθεια και εμείς βοηθάμε. Να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Συνεργάζονται άριστα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ε, συνεργάζονται ε, στα, ταξίδια που κάνουν και κινούνται και υπέρ των κρατών μελών, ο Κάρολ Μπίλ, ο Βίλιαν Χέμ κλπ. Ε, κάναμε μαζί ένα ταξίδι και θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Το θέμα των βοηθών. Πολύ σωστά είπατε ότι είναι αδύνατον ε, να είμαι πανταχού παρούσα. Εγώ θυμάμαι μια θλιβερή μέρα που πήγα σε πέντε χώρες σε μια μέρα και επεκρίθην διότι δεν πήγα στην έκτη χώρα. Είναι αδύνατον να πετύχει κανείς τα πάντα χωρίς να χρησιμοποιεί την πολυτιμότητα της υποστήριξη των διαφόρων προεδριών. Όταν όλα αυτά τα συναθρήσουμε όλες αυτές οι, προηγου... συνεδριάσεις που προηγούνταν πριν υπήρχαν. Τα συμβούλια σύνδεσης, όλα τα μορφώματα αυτά, οι τρόποι με τους οποίους συνεδριάζαμε. Αυτά με την πάροδο του χρόνου διαμορφώθηκαν, συνεχίστηκαν. Ε, παρόλα αυτά που ήταν ένα άτομο και όχι τρία. Έπρεπε να προεδρεύω τριών συμβουλίων. Οπότε η εναλλακτική προεδρία ήταν υπέροχη, διότι ε, επομίστηκε πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασία και ο Στέφαν Φούλερ το έκανε, συνεργάστηκα στενά μαζί του αλλά και άλλοι επίτροποι βοήθησαν. Ήταν πρόθυμοι να εκπροσωπήσουν εμένα και την Ένωση με διάφορους τρόπους και άλλοι και οι Υπουργοί Εξωτερικών βοήθησαν. Δεν είναι συνηθιστό να δείτε ότι ένας Υπουργό Εξωτερικών να κάνει μια ε, παρέμβαση για τη χώρα του κάνει και μια παρέμβαση εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι πολύ καλή χρήση των διαθεσίμων ε, πόρων και συστήνω αυτή τη μέθοδο δεν αφαιρεί τίποτα από το ευρύτερο, την ευρύτερη συζήτηση που απαιτείται, δηλαδή πώς αυτός ο ρόλος θα διαδραματιστεί, θα είναι ένα άτομο στο μέλλον, αν εξακολουθεί να είναι, να είναι πολλά τετήματα που βάλλονται και απαιτήσει για ένα άτομο. Τώρα το πώς εργαζόμαστε για τη διαχείριση των κρίσεων και την αποφυγή των συγκρούσεων πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα τη σφαιρική προσεγγίσεω. Πώ χρησιμοποιήσουμε τι επιδεξιότητε δημοσιολάβηση για την επιβολή κράτου δικαίου κλπ. Αυτά είναι σημαντικότατα ζητήματα και πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Και αυτό απαιτεί εξέταση. Να είμαστε σίγουροι ότι όλα ταιριάζουν μεταξύ του. Υπάρχουν διάφορε δομέ και έχουν εκκληρονομηθεί δομέ και εγώ δεν έχω και την εξουσία να τι αλλάξω. Μπορώ μέσω τη αναθεωρήσεω και με την υποστήριξη μάλλον τη δική σα και των κρατών μελών μπορώ να κάνω τι Παρομοίως, όταν σκεφτούμε και τη δουλειά που κάνουμε για την άμυνα και τις αποστολές της ΚΕΠΑ, δεν μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ ε, μακροχρόνιες, χρειάζονται πάρα πολλές επιτροπές για τη λήψη αποφάσεων κλπ. Αυτές οι σημαντικές αποφάσεις δεν προσπαθώ να τις μειώσω, δεν προσπαθώ να τις αφαιρέσω τα κράτη-μέλη, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να διατρέξουμε όλες τις διαδικασίες. Και κάτι που εισήγαγα, θα θυμόσαστε, ήταν στρατηγικές εξόδου, αλλά τις αποστολές δεν υπήρχαν, υπάρχουν. Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό εξαρτώμεθα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή τη δουλειά. Θα πρέπει να δούμε κάποιου κανονισμού που ισχύουν και χρειάζομαι τη βοήθειά σα γιατί χρειάζεται και χρειάζονται αρκετέ αλλαγέ. Μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συμφωνίας των θεσμικών οργάνων και μέσω αλλαγής κάποιων κανόνων και αλλαγής κάποιας νομοθεσίας. Αλλά πρέπει να γίνουμε ταχύτεροι και αυτό δεν θα συμβεί μόνο με ευχολόγια. Θα γίνει μόνο αν εμείς κάνουμε κάτι όσον αφορά τι πρεσβείε, αντιπροσωπείε κλπ. Αυτό που λέω ότι είναι ανοίγει πρεσβείε ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Βίλιαμ Χέγγ είναι πάρα πολύ περήφανο να σα πω εκ μέρου του ότι ανοίγουν και δεν κλείνουν πρεσβείε και προξενία. Υπάρχει και ένα ερώτημα που ετέθη για τα Μπαρμπέιτο ε, σε σύγκριση με τον Παναμά. Το Μπαρμπέιτο ε, δέχεται διάφορη αρνητική προβολή για λάθο λόγου. Θα εξηγήσω είναι κόμβο για περιφερειακή βοήθεια τα Μπαρμπέντο. Έχουμε 44 άτομα εκεί. Τρει είναι από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, έξι είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 35 είναι ντόπιοι. Και είναι για τη χορήγηση βοήθεια για 10 χώρε και εδάφη. Αντίγουα, Μπαρμπέιντο, Δομίνικα, Μπαρμπέιντο, Κιτσανέβη κλπ. κλπ. Είναι υπεύθυνοι για 250 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεων για τις χώρες. Αντί να έχουμε 10 διαφορετικούς τόπους με 10 διαφορετικές γραφειοκρατίες, τα μαζέψαμε όλα μαζί, αλλά είναι μόνο τρεις προσωπικό δικό μας. Οι υπόλοιποι χορηγούν αναπτυξιακή βοήθεια. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να, να ανοίξουμε και στον Παναμά και στον υπόλοιπο κόλπο και Στις χώρες του κόλπου. Πρέπει να το κάνουμε αυτό εν ευθέτω χρόνο. Χρειαζόμαστε όμως τους αναγκαίους ε, πόρους. Και αυτό είναι σημαντικό. Ανοίξαμε στη Λιβύη Ανοίξαμε στο Μιανμάρ, προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στι δραματικέ αλλαγέ, βάζοντα επιτόπου ανθρώπου που μπορούν να είναι παρόντε και να μείνουν εκεί. Αλλά αυτό κάθε αυτό είναι μια πρόκληση. Όσον αφορά τη στελέχωση, πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Κληρονομήσαμε, θυμηθείτε, περισσότερο, το περισσότερο προσωπικό από τα άλλα θεσμικά όργανα. Οπότε το φύλλο, το ιστορικό του, όλα αυτά κληρονομήθηκαν και η πείρα του. Και η αλλαγή σε οποιοδήποτε οργανισμό μα γίνει αυτό και έχω μεγάλη εμπειρία. Για να αλλάξει κάτι τέτοιο σαν οργανισμό χρειάζεται χρόνο. Πρέπει να δούμε ποιε διαδικασίε θα μπορέσουν να δώσουν δυνατότητα σε κόσμο να προσληφθεί. Προσπάθησα να φέρω περισσότερε γυναίκε στην υπηρεσία και χαίρομαι ότι έχει αυξηθεί αριθμό των γυναικών. Στα εθνικά διπλωματικά συστήματα δεν είναι τόσο πολλέ γυναίκε που αναμειγνύονται στην εξωτερική πολιτική. Θα πρέπει να επιλύσουμε λοιπόν κάποια προβλήματα, κάποια εμπόδια να έρθουν που υπάρχουν και το εξετάζουμε αυτό. Στέλνουμε κόσμο να πάει να μιλήσει με διάφορου πρωτεύουσε όπου υπάρχει υποεκπροσώπηση, να δούμε πώ θα πετύχουμε την ισορροπία. Δεν θέλω όμω να έχουμε ποσοστώσει. Θέλω βάση αξία να παίρνουν τη θέση του. Επικεφαλή αντιπροσωπεία ξέρει ο καθένα ότι πήρε τη δουλειά ή θεωρήσαμε ότι ήταν το καλύτερο άτομο για να εκπροσωπεί την Ένωση ε, και να κάνει τη δουλειά που απαιτείται να κάνουμε και ε, συμφωνώ και για, για τις διακοπές και του άλλους κανονισμούς. Δεν μπορούμε αν δεν αλλάξουμε τους κανονισμούς να αλλάξουν αυτά. Δεν έχει νόημα το πώς είναι η δομή για τις διακοπές και τι τις άδειες. Βέβαια, ε, κάποιοι σε δύσκολα πόστα χρειάζονται κάποιε διακοπέ. Κανεί δεν τα αμφισβητεί. Αλλά δεν βλέπω γιατί έχουμε διαφορετικέ ρυθμίσει. Ε, έτσι αναπτύχθηκε το θέμα. Αλλά για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει να αλλάξω τον κανονισμό. Άρα χρειάζομαι εσά. Αυτό αληθεύει και για άλλα πράγματα. Δεν είμαι κατά των αλλαγών. Αλλά ξέρετε και εγώ ξέρω ότι απαιτείται να κάνουν άλλοι προτάσεις και να υπάρξει συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι που απαιτεί κάποια προσεκτική αντιμετώπιση ευαισθητών θεμάτων. Οι προτάσεις που κάνουμε για τέτοιες αλλαγές λοιπόν έχουν υποβληθεί από τις ίδιες αντιπροσωπίες. Τους ρώτησα, είπα στους εκπροσώπους τους, δώστε μας τις ιδέες σας, τι πρέπει να κάνουμε και να δράσουμε βάσει αυτών. Βέβαια, ε, Επίσης εξέτασα και το τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την μείωση των θέσεων των ανωτέρων στελεχών. Από την αρχή που δημιουργήθηκε η υπηρεσία ξέραμε ότι ήταν μια δομή που χρειαζόμαστε για να απογειωθούμε αν θέλετε. Πρέπει να το επανεξετάσουμε. Πρότεινα να μειωθούν οι, ε, οι 6 αδ 16 και 9 αδ 15 για του χρόνου και πρότεινα στα κράτη-μέλη ε, να κάνουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τους ειδικού εκπροσώπους, να δούμε τι εντολές έχουν, να δούμε τι αριθμοί υπάρχουν και να δούμε πώς μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στην υπηρεσία αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό που είναι στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε καμιά φορά δυσκολότατες κρίσεις όπου χρειάζεται κάποιος ο οποίος δεν βρίσκεται με την έδα σε μια ε, περιοχή αλλά μπορεί να πάει και σε άλλα μέρη και καμιά φορά πρέπει να προωθούμε διάφορα ζητήματα που χρειάζεται συνδυασμό επικεφαλή αντιπροσωπεία και ευρύτερη εκπροσώπηση, όπω γίνεται στο Αφγανιστάν. Αλλά φέρνουν αυτοί οι άνθρωποι και προσωπικό που απαιτείται. Άρα όλα αυτά πώ θα ενταχθούν και θα ολοκληρωθούν ε, είναι το θέμα. Κανεί δεν είναι πιο αφοσιωμένο να, να το κάνει αυτό από μένα. Θέλω να το κάνω αυτό. Πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που θα εξασφαλίζει τη σωστή συνέχιση τη ανάπτυξή μα. Και τέλο, το θέμα αντιπροέδρου. Συμφωνώ συνομιλώντα με τον πρόεδρο Μπαρόσο, το, το, το, του τελευταίου μήνε συζητήσαμε. Συμφωνούμε, πρέπει να κάνουμε περισσότερο να τα αναπτύξουμε. Ε, το είπα στην αρχή. Έδωσα κάποια παραδείγματα πώ μπορούμε και συνεργαζόμαστε. Ε, με διάφορου επιτρόπου συνεργαζόμαστε για διαφορετικά ζητήματα. Αλλά συναντηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουμε για τη Συρία και για την άμυνα. Ξενθήκαμε του επιτρόπου και σε πολλέ άλλε περιστάσει μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Και ο πρόεδρο και εγώ Θέλουμε πράγματι να γίνουμε αποτελεσματικότεροι σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, σα ευχαριστώ ξανά κύριε Ευρωβουλευτέ για τη συζήτηση. Είπα πολύ συχνά ότι η δημιουργία τη υπηρεσία ήταν σαν να προσπαθήσει κανεί να απογειώσει ένα αεροπλάνο όταν ε, δεν έχουν μπει καλά-καλά τα φτερά και να φέρνουμε ε, στελέχια από άλλου χώρου και άλλα θεσμικά όργανα, από 7 διαφορετικέ τοποθεσίε από τι Βρυξέλλε και να του ζητούμε να δημιουργήσουν κάτι καινούριο και να ζητήσουν τι προσωπίε επιτόπου να υπομισθούν νέε ευθύνε χωρί του πόρου, Χρειάζονται βοήθεια όλα αυτά. Σε πόλεις όπως τη Νέα Υόρκη, όπου ήρθε η παρενέβη η Προεδρία, δώσαν άλλα 20 άτομα επί τόπου, παραπάνω άτομα. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Άρα προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται. Φιλοδοξία μου είναι, φτιάξαμε τα θεμέλια, είχαμε τρεις προτεραιότητες, είναι η γειτονιά μας εκεί που είμαστε, να αναπτύξουμε στρατηγική, στρατηγικές σχέσεις, το κάναμε και αυτό, και θέλουμε να οικοδομήσουμε τις αρχές της υπηρεσίας που μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να είστε περήφανοι για αυτή. Αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα να κάνουμε και με την υποστήριξή σας θα κλείσω εγώ τη θητεία μου και θα παραδώσω σκητάλη σε κάποιον άλλον τις αρχές ε, από κάτι που μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Και τώρα οι συγητές και πρώτα απ' όλα ο κύριος Ελμαρ Μπρόκ έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει δείξει ότι είναι πρόθυμο να, συμβάλλει στη βελτίωση της υπηρεσίας. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι αυτό κατεδείχθη με σαφήνεια στη συζήτηση που έγινε. Και περιμένω από εσάς ε, στην τοποθέτησή σας, ε, όχι βέβαια μια πλήρη απάντηση, γιατί νομίζω ότι τους επόμενους μήνες πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα θέματα που μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Και στο τέλος είπατε κάτι για τους κανονισμούς. Εκεί εντάσσεται και ο δημοσιονομικός κανονισμός και υπάρχουν και θέματα που πρέπει να τα αλλάξει ο νομοθέτης για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ε, και νομίζω ότι με την Κομισιόν και το Συμβούλιο θα τα καταφέρουμε. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν κάποια ωφέλη. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα που τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά να εμποδίζει τις ε, άλλες χώρες να δεχθούν τα προξενία. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και τον πολίτη. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να να τα εξετάσουμε γιατί από εκεί μπορούν να προκύψουν εξοικονομήσεις κοντιλίων για τα κράτη-μέλη. Το θέμα δεν είναι τι θέλει κανεί να κάνει αλλά τι μπορεί να κάνει. Όσον αφορά επίση του πολιτικού εκπροσώπου, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε αλλά θα πρέπει να συζητάσουμε, συζητήσουμε για το πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τον θεσμό των πολιτικών εκπροσώπων. Με άλλα λόγια, χαίρομαι για τι συζητήσει που θα ακολουθήσουν του επόμενου μήνε, Χαίρομαι για την εισήγησή σα, έτσι ώστε ώστε α, τον τελευταίο χρόνο αυτής της θητείας να μπορέσουμε να τον εκμεταλλευτούμε. Σας... Ο συνάδελφος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Grazie. Ma questo dibattito ha dimostrato, penso... Νομίζω αυτή η συζήτηση κατέδειξε ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη γραμμή της εκθεσής μας. Και με μεγάλη μου χαρά να ακούσω την άποψη του κυρίου Τάνοκ, ο οποίος θα αναφερθεί στο πόσο σημαντική είναι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Επίσης, η συζήτηση έδειξε ότι υπάρχει μια σημαντική σύγκληση ανάμεσα σε εσά και σε εσά, ε, κυρία Υπατή εκπρόσωπο. Κυρία Αστόν, μια θαυμάσια σε συζήτηση και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ όχι μόνο για ε, τις, ε, τα φιλοφρονήματα, τις φιλοφρονήσεις που επιδαψιλεύσατε στο Κοινοβούλιο αλλά και διότι καταδείξατε τις δυνατότητες που έχει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης απόψεις τις οποίες συμμεριζόμαστε εμείς πλήρως. Και χαίρομαι που αναφερθήκατε κυρίως ε, στην πρόκληση κατά τους επόμενους μήνες άρα δηλαδή και στη δυνατότητα να υπάρχει συνεργασία στα διάφορα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Ευρώπη για να μπορέσει να καταστήσει αποτελεσματική την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, έχουμε λοιπόν περιπτώσεις πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή. Τις περιπτώσεις αυτές τις υπενθυμίσατε. Υπάρχουν σαφώς αυτές οι επιπτώσεις. Θέλουμε βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτό τον τομέα υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά. Είμαι, ε, ε, ε, έχω εμπιστοσύνη ότι θα έχουμε μια πολύ καλή βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις. Είμαι αισιόδοξο και γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ εσά ε, και του ε, συνεργάτε σα ε, που βεβαίω ξεκινάω με τον κύριο Βιβμό για τη στράτευσή του, για τα αποτελέσματα που έχουν παρουσιάσει και για τη διαθεσιμότητα που είχαν πάντα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία για την έκθεση Μπροκ Γουαλτιέρη θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι κοινή συζήτηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα τη δημοκρατία